Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε γιατί στις 10 έχουμε και ψηφοφορίες. Μαζί μας σήμερα το πρωί είναι ο Υπουργός Ριμάντα Σινκεβίτσιους, Λιθουανός Υπουργός Μεταφορών και Συγκοινωνιών, εκ μέρους της Προεδρίας του Συμβουλίου. Θα είναι εδώ για τα επόμενα 40 λεπτά. Να τον καλωσορίσω λοιπόν. Ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε έξι πολύ δραστήριους μήνες, κάτι το οποίο θεωρώ βέβαιο. Εμείς ως Επιτροπή Ήτρε θα μεταβούμε στην Λιθουανία την επόμενη Δευτέρα, επομένως θα γίνει και μία πρώτη ε, συνάντηση στη χώρα σας. Ε, σας καλωσορίζω λοιπόν κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Λιφωνικής Προεδρίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους προκατόχους μας, την Ιρλανδική Προεδρία και πιο συγκεκριμένα τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ράμπιτ και την ομάδα του, ο οποίος με την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή σας ε, κατάφερε να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο σε θέματα τα οποία ενδιαφέρουν όλη την Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε, η Λιθουανία είναι η πρώτη από τις τρεις χώρες της Βαλτικής που αναλαμβάνει καθήκοντα Προεδρίας ε, του Συμβουλίου. Μάλιστα, λιγότερο από Δέκα χρόνια πριν, το 2004, υπήρξε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην ιστορία της χώρας μας όταν η Λιθουανία έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Λιθουανία θα προσπαθήσει να διασφαλίσει μια σταθερή και συνεχή νομοθετική διαδικασία σε μια διαδικασία που θα περιλαμβάνει τους πάντες αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδίως μετά την συνθήκη της Λισαβόνας, και στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα προσπαθήσουμε να έχουμε επικοδομητικές, αποτελεσματικές ε, και ε, αμοιβαία ε, συνεργασία με την Επιτροπή σας κυρίως οι προσπάθειάς μας θα επικεντρωθούν σε δράσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και των χρηματοπιστωτικών αγορών. Επιπλέον θέλουμε χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιο παράδειγμα ασφάλειας ε, και ε, ευημερίας. Στη διάρκεια της Προεδρίας θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια αξιόπιστη, ε, ανοιχτή και αποτελεσματική Ευρώπη. Όπως γνωρίζουμε η Λιθουανική, Ιταλική και Ελληνική Προεδρία θα είναι η ε, το τρίο το οποίο θα συνεργαστεί, η τελευταία προεδρία που θα συνεργαστεί με την παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην παρούσα θητεία, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αρκετά θέματα και να αποφασίσουμε επί αρκετών θεμάτων. Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας ε, στην, στο των Προεδριών για να διασφαλίσουμε συνέχεια και τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τώρα, θα πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη, ε, ε, ολοένα αναπτυσσόμενη και ανοιχτή Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια δυναμική, ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά. Να σας δώσω ένα διάγραμμα των όσων σκοπεύουμε να κάνουμε στο μέλλον. Καταρχάς, θέλουμε να έχουμε έγκαιρη συμφωνία και από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές του Διευρωπαϊκού Δικτύου Τηλεπικοινωνιών. Το επικαιροποιημένο κείμενο των ε, κατευθυντηριών γραμμών TEN Tele παρουσιάστηκε το, στα τέλη Μαΐου και σήμερα η Επιτροπή σας θα ψηφίσει επί του ζητήματος αυτού. Με χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχει σύμπνη απόψεων στο θέμα αυτών και ελπίζω μετά από τη σημερινή ψηφοφορία να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή σας τον κύριο Τοζενόφσκι, ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια βάση για ασφαλή, αξιόπιστη και εύκολη επικοινωνία μέσω διαδικτύου και συναλλαγές μέσω διαδικτύου, γεγονός το οποίο θα δώσει μια νέα όθηση στην αγορά των ηλεκτρονικών ε, υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν ε, διευκρίνησα στους Υπουργούς ε, στο Συμβούλιο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας του Ιουνίου ότι ο κανονισμός για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις ε, υπηρεσίες οι οποίες θα είναι αξιόπιστες αποτελεί προτεραιότητα για μας. Βεβαίως είναι αυτονόητο ότι πολλά πράγματα ακόμα εκκρεμούν προκειμένου να μπορέσουμε να επιλύσουμε πολύ σημαντικά θέματα τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πρόταση, ιδίως όσον αφορά το σεβασμό των αρχών της αξιοπιστίας, της εμπιστοσύνης και της διαλειτουργικότητας. Ελπίζω λοιπόν ότι η συνεργασία με τον εισηγητή σας την κυρία Μαρίτα Ούλσκοπ ε, θα είναι αποτελεσματική και θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια ε, θετική και επιδημοτική διαδικασία διαλόγου σε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Θα διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πρόοδο στο Συμβούλιο μέχρι να πρέπει να ψηφίσει η Επιτροπή σας για την πρόταση αυτή το Σεπτέμβριο. Προβλέπουμε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο στη διάρκεια της Προεδρίας μας και πάλι, με στόχο και πάλι να έχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Παραβίαση ηλεκτρονικού χώρου. Αυτή είναι μια ε, ταχύτατα αναπτυσσόμενη απειλή η οποία εξαπλώνεται πέραν του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Γίνονται προσπάθειες για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η απειλή και πρέπει να ληφθούν και αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ψηφιακή μας οικονομία και να έχουμε υγιή και αξιόπιστα δίκτυα και κατάλληλες ε, εγκαταστάσεις και υποδομές ε, ε, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Γι' αυτό ακριβώς και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε προοδό στην πρόταση για την οδηγία για τα δίκτυα και την ασφάλεια των πληροφοριών, να εντοπίσουμε τους βασικούς κινδύνους, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή ασφάλεια. Θα προσπαθήσουμε επίσης να επιτύχουμε πρόοδο στο Συμβούλιο στην πρόταση για τον κανονισμό για τα μέτρα για τη μείωση του κόστους ε, των ε, δικτύων ε, επικοινωνιών ε, ε, ευρυζωνικών προκειμένου να μειώσουμε το κόστος της υψηλής ταχύτητας επικοινωνίας σε ευρυζωνικά δίκτυα και να βελτιώσουμε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών για να υπάρχει ε, πραγματικά καθολική πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες να προσφέρουμε ε, διαδικτυακές υπηρεσίες και σε άτομα με αναπηρία. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να προχωρήσουμε και την οδηγία για την ε, πρόσβαση ε, των, σε ιστότοπους φορέων του δημοσίου τομέα. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε και τους στόχους ανάπτυξης του Ευρώπη 2020 θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και τον κανονισμό για τον οργανισμό για το ευρωπαϊκό ε, σύστημα ε, GPS και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι πρέπει να ε, έχουμε μια κοινή προσέγγιση στο Συμβούλιο, κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να επιτύχει η Προεδρία και θέλουμε να συνεργαστούμε και μαζί σας κυρία Πρόεδρε γιατί είστε η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συνεργασία μας για το θέμα αυτό. Είμαστε εν αναμονή και τη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή ευρωπαϊκή αγορά για τι τηλεπικοινωνίε. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους στόχους της πρότασης και τα κύρια προσκόμματα τα οποία θα πρέπει να υπερκεράσουμε προκειμένου να έχουμε μια σταθερή κοινή ενιαία ψηφιακή αγορά και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη και τα θέματα τα οποία ε, προέκυψαν στο ε, Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών του Ιουνίου. Οι συζητήσεις μεταξύ των Υπουργών αναμένεται να δημιουργήσουν μια πολύ σημαντική συνεισφορά στις συζητήσεις που θα κάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο, προκειμένου να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι η ψηφιακή ατζέντα για την ε, ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τη σχέση που έχει με την πολιτική καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Λιθουανία θα διοργανώσει το τη διάσκεψη ICT 2013 στο Βίλνιο στο Νοέμβριο. Αυτή η πολύ μεγάλη διάσκεψη θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Ε, και περιμένουμε να ε, επιδείξετε κι εσεί ανάλογο ενδιαφέρον, όπω και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι για τη διάσκεψη αυτή. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι ελπίζουμε να έχουμε έναν επικοδομητικό και φιλικό διάλογο, όπω ε, ξεκινάμε τις εργασίες μα για αυτό το τόσο σημαντικό θεματολόγιο. Ε, ο στόχο είναι κοινό, μια αξιόπιστη και ανοιχτή Ευρώπη και προσβλέπω στη συνεργασία για να επιτύχουμε από κοινού αυτό το στόχο. Σα ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ. Σας ε- θα έχουμε τις παρεμβάσεις, τις πρώτες παρεμβάσεις. Η κυρία Πιλάρ Καστίγιο, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο πλαίσιο της Επιτροπής Βιομηχανίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντική συνεργασία μαζί μας, αλλά ελπίζω να νιώθετε ότι εδώ θα είναι και το δεύτερο σπίτι σας κάθε φορά που θα έρχεστε στην Επιτροπή μας ή θα ήρθετε σε επαφή μαζί μας. Καλώς ορίσατε λοιπόν. Μας κάνατε μια πλήρω η επισκόπηση των θεμάτων τα οποία κρεμούν αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να σας πω ότι από τα θέματα ε, τα οποία άπτονται αυτές τις επιτροπές, τα οποία είναι πάρα πολύ ευρεία στην έκτασή τους. Ε, η βιομηχανία, η τηλεπικοινωνία, ε, τεχνολογίες πληροφορικής. Ο συγκεκριμένο τομέας, ο τομέας ε, για τον οποίο είστε αρμόδιος εσείς στη διάρκεια της ηλεκτρονικής προεδρίας, είναι ο τομέας ο οποίος είναι πιο δραστήριος στα τέλη αυτής της θητείας. και ελπίζουμε η Αντιπρόοδος ε, Νέλη Κρούς ε, με κάποιο τρόπο να ε, διατυπώσει όλα αυτά τα οποία μας έχει ανακοινώσει και να προχωρήσουν αυτά τα θέματα ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα μέχρι το τέλος της θητείας. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα όπως το θέμα της ηλεκτρονικής ταυτότητας και οι ασφαλείς υπηρεσίες υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε όπως ε, είπατε και εσείς ε, τα οποία αφορούν και την Επιτροπή μας όπως για παράδειγμα τις δορυφορικές υπηρεσίες και υπάρχει και ούτε λίγο το πολύ η οδηγία για τα ασφαλή δίκτυα. Θέματα λοιπόν κυβερνοασφάλειας τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν προεξάρχουσα θέση παγκοσμίω, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όσα κάνει η, Ευρωπή, η Επιτροπή μας εδώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ ευρύ θεματολόγιο και μη νομοθετικά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, συζητάμε το θέμα του cloud computing για να δούμε τι στάση θα τηρήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ναι, μεν αυτό το θέμα δεν είναι νομοθετικό, αλλά είναι λίγο ε, πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, διότι χαράσει λίγο την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε και υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα τέτοια φύσεω, τα οποία ναι, μεν δεν είναι νομοθετικά, αλλά είναι εξίσου σημαντικά. Να επικεντρωθούμε όμως στα νομοθετικά ζητήματα, το είπατε κι εσείς, για τα θέματα της ηλεκτρονικής ταυτότητας ε, και της ασφαλής υπηρεσίας. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά σύντομα, διότι ε, μέχρι του έχουμε διαπιστώσει εδώ στην Επιτροπή μας ότι υπάρχει αξιοσημείωτη ταύτιση απόψεων. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία εδώ στην Επιτροπή και δεν θα είναι δύσκολο να υπάρχει μια συνεκτική απόφαση ε, στο θέμα αυτό, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε και το θέμα αυτό σε πρώτη ανάγνωση. Τώρα, το θέμα της κυβερνοασφάλειας, ε, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι λίγο πιο περίπλοκο, διότι πραγματικά Νομίζω ότι είναι λίγες οι πιθανότητε να καταλήξουμε σε κάτι στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ο στόχο είναι να μπορέσουμε να το υπερψηφίσουμε στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο. Επομένως το λογικό θα ήταν αυτό, διότι είναι δύο ε, αρμόδιες, ε, δύο επιτροπές αρμόδιες. Ε, η επιτροπή μας ε, είναι μία εξ αυτών. Αλλά επειδή ούτω ή άλλω εσεί θα έχετε τα ενία τη Προεδρία, εγώ ζητάω την υποστήριξή σα και τώρα, αλλά και μετά, αφού θα έχετε ε, παραδώσει τα ενία σε άλλου και θα είστε απλώ μέλο του Συμβουλίου. Θα ήθελα να σας ε, θέσω κάποιες ερωτήσεις. Το ένα βέβαια το απαντήσατε ήδη. δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα μας παρουσιάσει η Αντιπρόεδρος ε, Νέλη σήμερα το απόγευμα, αλλά και εσείς είπατε ότι επιθυμείτε ο κανονισμός να περατωθεί το συντομότερο δυνατό και φυσικά και εσείς να μπορέσετε ως λεθουανική Προεδρία να βοηθήσετε. Από ό,τι βλέπω είναι θετική η στάση σας. Εγώ θα είμαι στο Βίλνιους ε, στη διάσκεψη ε, την οποία θα κάνετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ε, παρά το γεγονός ότι ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε και στη διάρκεια της δικής σας προεδρίας και στην επόμενη, ελπίζω ότι θα διαδραματίσετε ένα σημαντικό ρόλο και θα μπορέσετε να επιταχύνετε λίγο τις ε, διαδικασίες. Και ένα τελευταίο ζήτημα και με αυτό ολοκληρώνω και μια παράκληση. Το φθινόπωρο θα γίνει ένα συμβούλιο το οποίο θα ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά θα ασχοληθεί με την ψηφιακή αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ψηφιακό θεματολόγιο, το οποίο φυσικά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ψηφιακή αγορά και ε, αντιστρόφως φυσικά, αναλόγως με το ποιο πρίσμα εξετάζει ο καθένας τα θέματα και η Επιτροπή μας σε μία ώρα ε, περίπου θα ψηφίσει ένα ψήφισμα για το ψηφιακό θεματολόγιο και το μέλλον του ψηφιακού θεματολογίου. Ο τίτλος ε, λέει πολλά. Λέει ψηφιακή ατζέντα, άνω κάτω τελεία, ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Και έχει και έναν υπότιτλο. Στα αγγλικά λέει It's time to move up a gear, δηλαδή η η ώρα να επιταχύνουμε λίγο τα πράγματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η φωνή του Κοινοβουλίου, γιατί αυτό θα ε, ψηφιστεί πριν από τον Οκτώβριο, θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο, να φτάσει ε, μέχρι το Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θεωρούμε προτεραιότητα. Το θέμα της περιαγωγής, για παράδειγμα, το οποίο επισημαίνεται εδώ. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από πολύ ε, σημαντικούς τομείς ε, που επήγει να παρέμβουμε. Το ένα έχει σχέση με τις υποδομές, το δεύτερο έχει σχέση με την ανάπτυξη και την απασχόληση και υπάρχουν και άλλοι δύο τομείς οι οποίοι κατά την άποψή μου ε, είναι πολύ σημαντικοί, η πλήρης ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ψηφιακό τομέα. Θεωρώ ότι θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου όταν θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Κατά τα λοιπά, πραγματικά ελπίζω να νιώθετε εδώ σαν το δεύτερό σας σπίτι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ε, συναντώ εδώ και ελπίζω να σας ξανασυναντήσω σύντομα. Ευχαριστώ Πιλάρ, ο κύριος Ντοζανόφσκι από την UCR. Ε, κυρία Πρόεδρε, καλώς, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Είμαι ακόμα πιο ευτυχής που βρίσκεστε εδώ, γιατί σήμερα θα ψηφίσουμε μια έκθεση στον τομέα του διαδικτύου, στον τομέα των ψηφιακών. Είναι λοιπόν μεγάλη μας ευχαρίστηση που σας υποδεχόμαστε εδώ, αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι πεπισμένος, όπως και εσείς, ότι το διαδίκτυο ε, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο γιατί παρέχει τεράστιες δυνατότητες σε πολλαπλούς τομείς, ε, τον κοινωνικό, τον οικονομικό. Έχει μεγάλη σημασία για την ικανότητα της Ευρώπης ε, να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σημασία της έκθεσης που θα ψηφιστεί σήμερα από την Επιτροπή μας ε, ε, συνδέεται ή μάλλον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου πακέτου για δημοσιονομικούς λόγους ε, τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκαν στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ φορά τη χρηματοδότηση, οπότε πρέπει να ανασυντάξουμε όλα αυτά τα προγράμματα και να προσανατολιστούμε προς το ψηφιακό ε, θεματολόγιο, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε στενά για όλα αυτά τα θέματα. Μας ικανοποιεί ιδιαιτέρως που κατά την Προεδρία σας θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, εργασίες που εξελίσσονται πάνω από δύο χρόνια τώρα και θα θέλαμε από κοινού να οριστικοποιήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, μάλλον τον Οκτώβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν τα κείμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσουμε επιτέλους να κλείσουμε αυτό το θεματολόγιο. Ε, κύριε Υπουργέ, ε, μία ερώτηση λίγο ευαίσθητη. Ε, έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι έχετε λίγα μέσα στη διάθεσή σας σε σχέση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να στηρίξουμε τις τεχνολογίες εχμής, ε, δεδομένης και της κατάστασης της οικονομίας που μας δίνει περιορισμένα οικονομικά μέσα. Οπότε το εγχείρημα γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Ε, τι, τι σκέφτεστε, ποιες ιδέες έχετε, θα μπορέσουμε το φθινόπωρο να αυξήσουμε ίσως τα χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας για να εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους. Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας. Πώς βλέπετε την δυνατότητα ε, μιας ταχύτερης ε, οικονομικής, ε, μιας ταχύτερης τεχνολογικής εξέλιξης. Ανυπομονώ τον να έρθει ο Οκτώβρης και να συνεργαστούμε από κοινού και με τους άλλους εταίρους μας μετά μετά από δύο χρόνια που πέρασαν είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε αυτό το καθήκον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Κοτσανόφσκι. Παλιτσίτης. Ε, Κύριε Πρόεδρε, δράτω με τις ευκαιρίες για να Καλώς και εγώ τον Υπουργό. Τον Υπουργό Σενκεβίτσιους τον ξέρω πολλά χρόνια και είμαι σίγουρος ότι είναι εξαιρετικός ε, στη δουλειά του, είναι πολύ έμπειρος. Γνωρίζει πολύ καλά τους διάφορους τομείς και τα θέματα και είμαι σίγουρος ότι η Προεδρία σε των τον τομέα θα είναι επιτυχής. Το ψηφιακό θεματολόγιο είναι ένα τμήμα των εργασιών της δικής μας Επιτροπής γιατί μιλούμε για ένα πολύ ευρύ κλάδο ευθυνών αρμοδιοτήτων. Η κυρία Δελκαστήγιο μίλησε για τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ατζέντα. Δεν θα ήθελα λοιπόν να τα επαναλάβω. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι η Λιθουανία θα προσπαθήσει να ενισχύσει την αγορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και να ενθαρρύνει την περαιτέρω εξέλιξή της. Βεβαίως πολλά εξαρτώνται από την ηλεκτρονική υπογραφή. Το θέμα αυτό ακόμη εκρεμεί σε πολλές χώρες. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω τη δική σας άποψη, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να υπάρξει πρόοδος το τομέα. Τέλος, να σας ευχηθώ κάθε καλό, κάθε επιτυχία στην ομάδα σας και σε εσάς. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρετε και θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο E Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Πιστεύω ότι η Προεδρία σας θα είναι σημαντική ε, τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και των τηλεπικοινωνιών. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας των τηλεπικοινωνιών. Ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή νιώθουμε ότι απειλείται τόσο από τον κυβερνοασφάλεια, δηλαδή την παρίσφρηση στις τηλεπικοινωνίες άλλων στοιχείων, αλλά ε, και για πολύ πιο περίπλοκα, περίπλοκες παραμέτρους που καθίστανται τεχνολογικά εφικτές και θα ήθελα πολύ αυτά να βρουν μια παρουσία στην ευρωπαϊκή πολιτική. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω την δυνατότητα να έχουν παρισφρήσει κυκλώματα τα οποία είναι σε θέση να αντιδρούν σε λέξεις κλειδιά και να μεταδίδουν το περιεχόμενο των δικών μας συνομιλιών και δραστηριοτήτων για σκοπούς, ή για σκοπούς ε, πολύ ευαίσθητους από άποψη κατασκοπίας. Κάτι που θα ήθελα να ζητήσω συγκεκριμένα θα ήταν να ε, έστω και σε στατιστικό επίπεδο να γίνεται ένα συνεχής έλεγχος έτσι ώστε να διασφαλιστεί ένα καλό επίπεδο ασφάλειας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να απειλούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στις διαστημικές επικοινωνίες, δηλαδή στο δορυφορικό δίκτυο ε, στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών. Γνωρίζετε τους κινδύνους ε, υπάρχει καταρχήν ένας κίνδυνος σύγκρουσης με τα διαστημικά απορρίμματα όπως τα αποκαλούμε. Και επίσης υπάρχουν οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις ηλιακές θύελες. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ζητήσω να επιδείξετε μεγάλη επιμέλεια έτσι ώστε αυτά να ενταχθούν στην έρευνα και την τεχνολογία λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι υποδομές είναι πραγματικά ευρωπαϊκές και θα ήταν σκόπιμο να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει φυσικά να υπάρξει και μια χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι οι υποδομές αυτές θα τα πληρωθούν στο προσεχές μέλλον και δεν πρέπει να φοβόμαστε, ιδίως ε, εν μέσω της κρίσης, να επενδύσουμε σε αυτές τις ευρωπαϊκές υποδομές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφε Πρόντι. Δεν έχουν ζητήσει άλλοι τον λόγο. Σας δίνω λοιπόν κύριε Υπουργέ τον λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χάρηκα πολύ με τις ε, εξειδικευμένες απόψεις των μελών της Επιτροπής αυτής, ειδικά σε ό,τι αφορά τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η κυρία Πιλάρδελ Καστίγιο ανέφερε πολύ ευρεία κλίμακο θέματα που συζητώνται στην Επιτροπή σας. Ε, βλέπω ότι είσαστε λοιπόν πολύ εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό. Είπατε ότι ε, η θητεία όντως ε, ολοκληρώνεται και η ε, Λιθουανία θα προεδρεύσει για 4,5 μήνες περίπου γιατί το καλοκαίρι θα γίνει και ένα σχετικό διάλειμμα και εσείς το χρειάζεστε και εμείς. Μιλήσατε για την ε, εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία των ε, ε, ηλεκτρονικών αγορών, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την ηλεκτρονική υπογραφή. Όλα αυτά βρίσκονται στην ατζέντα μας, θα τα συζητήσουμε βεβαίως και μαζί σας και με τα υπόλοιπα 28 κράτη-μέλη. Ο κύριος Στοσενόφσκι μίλησε για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να μειώσει τον ε, προπολογισμό από 9,2 δις σε 1 δις για τις τηλεπικοινωνίες. Παρ' όλα αυτά, οι κατευθυντήρες γραμμές για τις τηλεπικοινωνίες έχουν ε, πραγματικά πολύ μεγάλο δυναμικό σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξη της οικονομίας. Και αυτό είναι νομίζω η ουσία του ψηφιακού θεματολογίου. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει, θα υπάρξει εφαρμογή των ε, κατευθυντήριων να πρέπει να συζητήσουμε μαζί. Ελπίζω λοιπόν ότι τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική απόφαση. Ο κύριος Μπαλτσίτης έθεσε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σχετικά με την ε, ε, περαιτέρω ανάπτυξη της ε, ενίας αγοράς, ε, την ηλεκτρονική υπογραφή και την αναγνώριση αυτής, καθώς επίσης και, τις, και το τι θα κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Η πρόταση αυτή είναι ιδιαίτερος περίπλοκη, αλλά για την ηλεκτρονική Προεδρία αποτελεί προτεραιότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά που ξεκίνησε η Ιρλανδική Προεδρία στον τομέα αυτό. Θα προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε, να συγκεράσουμε τις απόψεις των κρατών μελών και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια θέση του Συμβουλίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε συνεργασία, σε συζητήσεις, σε διάλογο με το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο στο θέμα αυτό, το συντομότερο δυνατόν και καλωσορίζουμε βεβαίως το γεγονός ότι η δική σας Επιτροπή έχει σκοπό να ψηφίσει ήδη για το θέμα αυτό από τον Σεπτέμβριο. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για, την, ε, ε, για τα καλά σας λόγια και για τις ευχές σας. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Πρόντι, μίλησε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο. Το θέμα αυτό όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό. και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μειώσουμε τις απειλές στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία, να υπάρχει εμπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στους σχετικούς παρόχους. Θα προσπαθήσουμε να επιφέρουμε πρόοδο και σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήρες γραμμές για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει όντως πρόεδρος, πρόοδος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως για την ε, πρώτη αυτή συνάντηση μεταξύ ημών και ημών που μας έδωσε τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και να κατανοήσουμε τι ακριβώς σκοπεύετε να προωθήσετε ε, στο διάρκεια αυτής, στη διάρκεια αυτής της εξάμενης συνεργασίας μας. Ε, ελπίζω να σας ξαναδώ εδώ σύντομα μαζί μας και εντωμεταξύ θα έχουμε σίγουρα τη δυνατότητα να συνεργαστούμε ε, και εμείς και με τους συναδέλφους ε, επί των θεμάτων που συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλή δουλειά. Bene, ora abbiamo 20 minuti. Ωραία λοιπόν. Έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Στις 10 να είστε όλοι εδώ για τη ψηφοφορία, διότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Διάλειμμα μέχρι στις 10. Bene, buongiorno. Proviamo. Καλημέρα. Για ελέγξτε όλη την κάρτα ψηφοφορία σας. Παρακαλώ να επαληθεύσουμε ότι λειτουργούν οι κάρτες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Μια στιγμή. Εντάξει. Πέρας της ψηφοφορίας. Έχουμε δύο πλεονάζοντες. Βγάζω λοιπόν τη δική μου κάρτα. Μία λιγότερη. Όλα εντάξει. Τέλεια. Ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτα έχουμε την έκθεση Μέρκης. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, ας κάνουμε μια επαλήθευση ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε δύο παραπάνω μέλη του Λαϊκού Κόμματος. Έβγαλα λοιπόν την κάρτα μου, άλλος ένας. Τέλεια. 26 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. Τούρμες υπέρ, κατά. Λοιπόν, επαλήθευση. Ψηφίζουμε την τροπολογία 16 τούρμες. Πέρας της ψηφοφορίας, 22 υπέρ, 27 κατά, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Α, επαλήθευση για την, την συμβιβαστική τροπολογία 28. Χολ. Πέρα της ψηφοφορίας. Πάλι έχουμε ένα πλεονάζον μέλλον του Λαϊκού Κόμματος. Ε, ένας βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος πρέπει να αφαιρέσει την κάρτα του. Εντάξει. Τέλεια. 46. Υπέρ 4. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική πρόταση 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αλλά θα κάνουμε επαλήθευση για την τροπολογία 35 το δεύτερο τμήμα πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία... Παρα... Ε, εντάξει, έλεγχος για την 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, πάλι έχουμε έναν παραπάνω βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος, αλλά δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. 26 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω πως έχει εγκριθεί. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας. Πάλι ένας παραπάνω βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος. Βγάλτε την κάρτα. Ωραία. 22 υπέρ, 29 κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Α, έλεγχος για την τροπολογία 60. Αρχίζει. Πέρας. 28 υπέρ, 23 κατά εγκρίνεται. Συγγνώμη, τουρμές. Συμβιβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 77. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, έλεγχος ηλεκτρονικός για την 77. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ένας επιπλέον βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος. εκτός μικροφώνη παρέμβαση ήταν 21 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. Ήταν... Για να δούμε... Τροπολογία 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Η πλειοψηφία κυμαίνεται πολύ σήμερα το πρωί. «23 υπέρ, 28 κατά». Απορρίπτεται. Τροπολογία 14, συμβιβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, αλλά... Ε, εγκρίνεται κατά τη γνώμη μου, αλλά ας επαληθεύσουμε. Με συγχωρείτε, αλλά ψηφίζετε πολύ λίγοι σήμερα το πρωί, πλειοψηφία κυμαίνεται και το βρίσκω δύσκολο να παρακολουθήσω. Τροπολογία 81 λοιπόν. 50 υπέρ. Ο, ο, ο, όλοι δηλαδή είχαν σηκώσει το χέρι. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, ελέγχουμε για την 82. Πέρας της ψηφοφορίας. 29 υπέρ, 21 κατά. 83 εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 24 κατά. Άρα απορρίπτεται. 24-24. Απορρίπτεται γιατί υπάρχει ισοψηφία. 21 υπέρ. Ο, με συγχωρείτε, λέει η πρόεδρος. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά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 Πέρας της ψηφοφορίας. «49 υπέρ και μία αποχή». Συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια. Προφορική ερώτηση. Εισηγητής υπέρ. Μια στιγμή. Ρόντε είναι ο εισηγητής. Αποχές ε, εγκρίνεται. Ψήφισμα Ρόντε. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας για την Ρόντε μάλλον τελική ψηφοφορία για την έκθεση Ρόντε. Πάλι ένα επιπλέον μέλος του Λαϊκού Κόμματος. Πέρας της ψηφοφορίας. 51 υπέρ. Συγχαρητήρια κύριε Ρόντε. Ας περάσουμε στην έκθεση το Ζανόφσκι. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Παρακαλώ. Η 21 και 22 καλύπτονται από την τροπολογία 1. Αν εγκριθεί 1 λοιπόν αρκεί. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 32 κατά τμήματα. Συγγνώμη 31. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 κατά τμήματα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 38, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 παρακαλώ. Μία επαλήθευση για τη 43. Παρακαλώ. Πέραση της ψηφοφορίας. Ένας επιπλέον από το ΕΛΚ. Εξακολουθεί. Ωραία. 30 υπέρ, 20 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ,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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, 70, ε, τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 8 υπέρ, επαλήθευση για την 7.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 Ψηφίζουμε για τις τροπολογίες υπέρ ηλεκτρονικά. Πρώτη ψηφοφορία λοιπόν για τις ε, τροπολογίες που εκρίθηκαν. Ένας επιπλέον από το ΕΛΚ. Πέρασε ψηφοφορία, 43 υπέρ, 6 αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το νομοθετικό ψήφισμα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 6 εποχέ. Ψηφίζουμε για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 50 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Τοζενόφσκι και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση του κυρίου Ρούμπικ. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Τροπολογία 42. Μπούτι κόφερ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 και 63 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ο συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 94 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 98 υπέρ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 Εξαιρετική η δουλειά σας. Έχουμε τώρα ένα προφορικό ζήτημα για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την προφορική ερώτηση. Πέραση της ψηφοφορίας. 51 υπέρ, καμία αποχή, καμία αρνητική ψήφους. Ευχαριστώ πολύ. Και πέρα της ψηφοφορία, λοιπόν. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν θα ξανακάνουμε ψηφοφορίες. Συγχαρητήρια λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, ζητώ συγγνώμη για το πρώτο τμήμα που ήταν λίγο περίπλοκο. Και τώρα κάνουμε τρία λεπτά διάλειμμα για να μπορούν να φύγουν από την αίθουσα όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν, ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια ήσυχα ήσυχα να κάνουμε τη δουλειά μας. Όλοι όσοι δεν θα παραμείνουν λοιπόν στην αίθουσα, παρακαλώ να αποχωρήσετε σε αυτό το διάστημα.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 Ας συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Μπιουτικόφερ, νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης για την προαγωγή της, της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας. Ο λόγος πάει στην κύριο Ράινχαρτ Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι κυρίως για τις δικές σας ε, απόψεις. Αυτές θέλω να ακούσω. Γι' αυτό θα είναι σύντομες οι δικές μου παρατηρήσεις. Ούτως ή άλλως η δική μου συμβολή στη συζήτηση θα είναι η γραπτή έκθεση. Αρχικώς να πω ότι έχουν συμπεριληφθεί σχεδόν όλα τα όσα μας έχετε προτείνει σε παλαιότερες συζητήσεις και μέσω παρατηρήσεών σας. Οπότε... Βέβαια δεν είναι όλα αυτά που γράφω εγώ, που γράφει η έκθεση μόνο δική μου ε, συγγραφή ε, προσπάθησα, δεν είναι μόνο δικές μου ιδέες, προσπάθησα να συμπεριλάβω και τα δικά σας σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας και γι' αυτό σας ευχαριστώ που μου τις στείλατε. Τώρα, η έκθεση αυτή ακολουθεί την ε, ανακοίνωση της Κομισιόν του προηγούμενου Οκτωβρίου. Ξεκινώ με κάποιους βασικούς στόχους και αρχές για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Βιομηχανίας και σε αυτή την ε, πρόταση εκθέσεως τονίζω και την σημασία που δίνει η Κομισιόν σε αυτή την πολιτική. Τονίζω την Ευρωπαϊκή Πολιτική Βιομηχανίας και όχι μόνο την ε, βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη θα το διαπιστώσετε αυτό και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου μιλούμε για βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ενσυνείδητα, όπως το προτείνει και η Κομισιόν, να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να μιλήσουμε για ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Αυτή είναι η διαφορά που βλέπω εγώ. Μιλούμε δηλαδή για έναν κοινό ορισμό στόχων και βασικών ε, αρχών. Σημαντικό επίσης είναι και νομίζω ότι θα ε, την χάνει αυτό και ευρεία ε, ε, συμφωνίας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να ακολουθήσει κοινού στόχου και επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για την προσέγγιση της, που έχει επιλέξει η Κομισιόν προς αυτό. Μια οριζόντια πολιτική δηλαδή. Όχι, δεν προσπάθησε να φτιάξει ξεχωριστου ε, πυλώνε, ε, ένα από τον οποίο να είναι η βιομηχανία όπω γινόταν στο παρελθόν. Τώρα έχει επιλέξει η Κομισιό να προχωρήσει με μια οριζόντια προσέγγιση, η οποία θέτει γενικώ το ερώτημα ποιε είναι, ποιες είναι οι ε, προποθέσει πλαίσιο μέσα στι οποίε πρέπει να λειτουργήσουμε, αν πρέπει να αλλάξουν ώστε να έχουμε μια, μια αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική, ώστε να δημιουργηθεί μια καλή βάση. Επίσης, Μιλούμε για την βιωσιμότητα, μιλούμε για την ανταγωνιστικότητα. Το αναφέρει και η Κομισιόν ρητά στην, στην ανακοίνωσή της. Μιλούμε για αναγέννηση της βιομηχανίας, για μια βιώσιμη Ευρώπη. Επίσης, ε, υπάρχει μια απόχρωση που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την ε, τεχνολογική ε, επίθεση ως προς την ε, εγκομηχάνηση. Επίσης, δίνεται μεγάλη σημασία στην εσωτερική αγορά. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα η οποία δεν έχει μόνο σχέση με τούτη την έκθεση, αλλά πάντα την έχουμε στο μυαλό μας, ότι πρέπει δηλαδή να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει έναν θεμελιώδη στόχο χωρίς την ενίσχυση της ιστορικής ε, εσωτερικής αγοράς δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους πολύ σωστούς στόχους που έχουμε θέσει αν δεν έχουμε μια σωστή, ένα σωστό μακροοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργούμε. Επίσης, σημαντική ε, σημασία δίνω και εγώ στην έκθεσή μου σε δύο πτυχές οι οποίες ε, μου τονίστηκαν ε, από πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, με τις, και στις συζητήσεις που είχαμε. Καταρχάς, το θέμα της πρόσβασης σε αξιόπιστη χρηματοδότηση. Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα ανά κράτος μέλος αλλά οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικώ βρίσκονται υποπίεση. Γι' αυτό εδώ κάνουμε κάποιες επιπλέον προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να γίνει, να διευκολυνθεί μια τέτοια πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι, σημαντικός, είναι ο τομέας των προσόντων και του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Και, αυτό είναι κάποιες, ε, και, ως προς αυτό έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, έτσι όπως το κάνει και η Κομισιόν στην ε, ανακοίνωσή της. Τέλος, δύο μικρά κεφάλαια έχω προσθέσει που θέλουν να τονίσουν λίγο περισσότερο δύο πράγματα. Ε, το ένα είναι μόνο τρεις παράγραφοι, παράγραφοι βέβαια, αλλά μιλούμε για τους πόρους και για την ενέργεια στο ένα κεφάλαιο. Νομίζω ότι αν ε, αυτό, που, αν δεν, αυτό παρόλο που δεν αναφέρεται ως συγκεκριμένος στόχος στην ανακοίνωση κομισιών, την βιομηχανική πολιτική δεν μπορούμε να τη συζητήσουμε ανεξάρτητα από το θέμα των πόρων και της ενέργειας. Και νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν σωστό να δούμε το θέμα ξεχωριστά και να του δώσουμε τη βαρύτητα που του αναλογεί, κυρίως για τις νότιες χώρες. έτσι ώστε να υπάρξει και εκεί μια βιομηχανική αναγέννηση. Να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλαν στις διάφορες συζητήσεις που κάναμε και βεβαίως περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ο λόγος των Προύστ. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή ε, για τη δουλειά του. Πριν απ' όλα, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στο σωστό πλαίσιο την αποστολή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ζητήσει τη γνώμη μας πάνω στο θέμα αυτό. Εμείς μόνοι μας σκύψαμε πάνω σε αυτή την προβληματική και, κατά το καν... και καλά κάναμε. Ε, είναι καλή αφετηρία η Επιτροπή μας, αλλά έχουμε περιορισμένη θητεία. Συχνά περιοριζόμαστε σε διαπιστώσεις, σε προβληματισμούς, αλλά δεν λαμβάνουμε πραγματικές δεσμεύσεις. Υπάρχει μια κρίση της βιομηχανίας αυτόν τον καιρό. Χρειάζονται απλά, καινοτόμα και συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό πρέπει να μας οδηγήσει στο να συμμεριστούμε τις ανησυχίες του κλάδου και να, να επιφέρουμε τις καλύτερες λύσεις. Αυτός πρέπει να είναι ε, ο στόχος μας, να δώσουμε απαντήσεις έτσι ώστε η βιομηχανία να ξαναβρει την ανταγωνιστικότητά της έτσι ώστε να έχουμε νέες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια πιο πράσινη βιομηχανία, αλλά προσοχή. Να μην είμαστε ιδεαλιστές, να μην ε, υποσχόμεθα μια επανάσταση βιομηχανική που θα είναι πιο πράσινη και θα δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας μέσα σε 12 μήνες. Προσοχή. Και με συγχωρείτε που θα πω, χρησιμοποιήσω αυτή τη συνηθισμένη φράση, να μην προτρέχουμε, να μην βάλουμε τα βόδια μπροστά από το άρωτρο πίσω από το μπροστά από το άρωτρο. Ε, πρέπει να ενσκύψουμε στο, στα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε μια κατάρρευση της βιομηχανίας. Ε, πρέπει δεν πρέπει να σκεφτόμαστε να διαμορφώσουμε την παραγωγή σύμφωνα με τις επιθυμίες μας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, τόσο για τη βαριά βιομηχανία, υπερπαραγωγή, όσο και για την κλάδο υψηλής τεχνολογίας μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού. Ανταγωνισμός διεθνής, γιατί σε άλλο τόνο, ε, σε ένα άλλο επίπεδο, Υπάρχει, είμαστε η πιο γυραιά βιομηχανική χώρα, βιομηχανική περιοχή στον κόσμο. Όμως ε, οι αναδυόμενες χώρες ε, έρχονται στο προσκήνιο ε, πολύ ορμητικά. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάποια πράγματα. Αν δεν κάνουμε τίποτα, αν μείνουμε αδρανείς, δεν θα επιβιώσουμε για πολύ καιρό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Δεν πρέπει τα κράτη-μέλη να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε τομείς που δεν έχουμε και καθόλου βιομηχανική παραγωγή. Σε τομείς που καλό θα ήταν να συνεργαστούμε όλοι, αν όχι να συγκλίνουμε ε, έχουμε τα θέματα της ποιότητας, το εργασιακό δίκαιο. Αυτά όλα πρέπει να τα διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τις βιομηχανίες μας, να τις συνοδεύσουμε, να τους βρούμε διέξοδο στις αγορές. Ε, η βιομηχανία μας χάνει όλο ένα και περισσότερο βάρος. Η Ευρώπη πρέπει να επανεκκινήσει την πορεία της βιομηχανίας της. Πρέπει να επιλέξουμε το δρόμο μας στον παγκόσμιο επίπεδο ως Ευρωπαίοι. Είτε είμαστε, ή είμαστε εταίροι, είτε είμαστε εταίροι, είτε είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε και το δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αν είμαστε εταίροι πρέπει να υπερβούμε τα σύνορα έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να μιλά με μία φωνή στον βιομηχανικό κόσμο. Γιατί το προβάδισμα δεν είναι πια στο εθνικό, αλλά στο παγκόσμιο επίπεδο. Τέλο, συμμερίζομαι τι απόψει του εισηγητή για την καινοτομία. Πρέπει να είμαστε στην καρδιά τη καινοτομία οι νέες τεχνολογίες θα μας φέρουν καινούργια πλεονεκτήματα ανταγωνιστικά. Έχουμε όμως μια αναπηρία στην Ευρώπη. Έχουμε εξαιρετική τεχνογνωσία, αλλά δεν την μεταδίδουμε στους άλλους. Πρέπει να συνοδεύσουμε τις επιχειρήσεις μας. Να, συχνά είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν τις καλύτερες ιδέες, αλλά δεν μπορούν να τις φέρουν στον ανταγωνισμό. Δεν ξέρουν ποιες πόρτες να χτυπήσουν. Νομίζω ότι δεν ανταποκρινόμαστε αρκετά γρήγορα και αρκετά ικανοποιητικά στις απαιτήσεις τους. Πρέπει να γίνουμε πιο φιλόξενοι στις επιχειρήσεις όπως η Ασία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, της Αμερικής. Πρέπει λοιπόν να συνοδεύσουμε καλύτερα, να διοχετεύσουμε τις χρηματοδοτήσεις μας πιο επιτυχώς, να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία και να διατηρήσουμε τα μυστικά μας για να προάγουμε την τεχνογνωσία και την καινοτομία μας. Πρέπει να συγχρηματοδοπτήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, πράγμα που δεν το συμμερίζεται μυστηριωδώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν οι άλλες χώρες. Ε, όπως την προαγωγή της, επιχειρηματι... της επιχειρηματικότητας διακινδύνευσης, τη διαπίστωση πιο ευνοϊκών μέσων χρηματοδότησης. Πολλές φορές ε, το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να παρέχουν αρκετές εγγύησεις στις τράπεζες για να τύχουν χρηματοδότησης. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν πρέπει να το ανοιχτούμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Κύριε Ανδρές Μπαρέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, βλέπουμε με πολύ θετικό τρόπο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ επίκαιρη και να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπουτικόφερ για την ε, ε, πρόταση που μας κάνει στο σχέδιο εξησής το οποίο βελτιώνει πολύ σημαντικά τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανεκβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν θα πρέπει να σταθούμε μόνο στην ε, βιομηχανική πτυχή, αλλά όπως είπε και ο κύριος Μπιουτικόφερ, θα πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκή πολιτική βιομηχανίας, αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να γίνει αναφορά σε θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την εκβιομηχάνηση της Ευρώπης, η ενέργεια, οι πρώτοι σόιλες, τα θέματα επιμελητίες ε, και θέματα ανταγωνιστικότητας και ε, βιομηχανίας. Η ανταγωνιστικότητα δεδομένου ότι έχουμε μία ένωση μεταξύ των νέων τεχνολογιών και της παραδοσιακής βιομηχανίας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τι αλληλεπίδραση και αγωνισμός υπάρχει μεταξύ κρατών μελών που αυτή τη στιγμή είναι ε, πολύ έντονος. Θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση, ισοδυναμία τίτλων θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση ε, μέσω προπολογισμού, διότι όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες παρουσιάζονται ως πολιτικές δράσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από κατάλληλο προϋπολογισμό και δημοσιονομικές προπτικές και πρόκειται και για μία έκθεση η οποία θέτει το θέμα της νέας ε, εκβιομηχάνησης της Ευρώπης ως διέξοδος από την κρίση. Υπάρχει μαζική έλλειψη θέσεων εργασίων σε αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, προτείνει μέτρα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή και πρέπει να το λύσουμε τώρα και να σχεδιάσουμε και πράγματα για το μέλλον. Αναμένουμε λοιπόν κατάλληλες πολιτικές και μέτρα όθησης τα οποία θα καταθέσουμε θέσουμε σε σχετικές τροπολογίες για να λάβουμε μέτρα βράχη πρόθεσμα, μέσο πρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Συγχαρητήρια και στον εισηγητή για την τοποθέτησή του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζόνσον. Γιώχανσον, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψει για, για το, το σχέδιο έκθεση και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με του προηγούμενου συναδέλφου που λένε ότι είναι καλό το γεγονό ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει τη σχετική έκθεση. Είναι κάτι που πρέπει και εμεί να μελετήσουμε και θα ευχαριστήσω και τον εισηγητή για τι προτάσει που έχει ήδη κάνει για τούτη την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πολύ καλέ οι προτάσει του. Αντιμετωπίζουμε όντω πολλέ προκλήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μιλούμε για βιομηχανικά θέματα, πολλές προκλήσεις λοιπόν και εδώ εμείς στην Ευρώπη πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις, προκλήσει. προκλήσεις. Δεν είμαστε σε ανταγωνισμό ένας με τον άλλον, πρέπει να, να συντονιστούμε μεταξύ μας, να συνεργαστούμε μεταξύ μας και αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει και εντός της Ευρώπης αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε την ενιαία μας αγορά, να γίνει αυτό βεβαίω με διαφανή τρόπο έτσι ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί στο μέλλον και αυτό είναι μία, αυτή είναι μία από τι πτυχέ που με ενδιαφέρουν εμένα. Θέλω να δω περαιτέρω δυνατότητε για ενοποίηση, για άνοιγμα τη εσωτερική μα αγορά. Έχουμε κάποιε επιμέρου αγορέ, δηλαδή κάποιε γεωγραφικέ αγορέ στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και μία ευρωπαϊκή προοπτική και θέλω και τι δύο να τι δούμε. Μιλούμε για πάνω από 500 εκατομμύρια πολιτών στο τέλος τέλος. Είναι πολύ καλό που έχουμε μια τέτοια πλατφόρμα και πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα έτσι ώστε να είμαστε και στη διεθνή σκακέρα πιο δυνατοί παίχτες. Πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε την αγορά μας, πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα για την αγορά μας και γι' αυτό χρειάζονται πολλές πρωτοβουλίες, όπως το Connecting Europe. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να εξασφαλίσουμε ότι οι υποδομές θα βελτιωθούν, ότι θα βελτιωθούν οι ευκαιρίες που δίνονται, θα, το, δούμε τον τομέα των μεταφορών ή τη ενέργεια. και εκεί θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Επίσης, υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, το δυναμικό των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ ε, πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, πολλές ευκαιρίες για καινοτομία και επίσης υπάρχουν και δυνατότητες για να υπάρξει όντως αυτή η αναγέννηση της βιομηχάνησης, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να αναγεννηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε και τον ορίζοντα 2020, εκεί χρησιμοποιούμε και τα, και τα clusters. Νομίζω ότι είναι και αυτά κάποια καλά εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση του εισηγητού, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το εμπλουτίσουμε λίγο παραπάνω με περισσότερε προτάσει. Ξέρω βέβαια ότι μπορεί να μην είναι θέμα ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά το θέμα τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι τομεί στου οποίου μπορούμε να δράσουμε περισσότερο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Τα συστήματα εκπαίδευση και κατάρτιση θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ περισσότερο και να ενσωματώσουν του πολίτε πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνουν τώρα. Κλείνοντα, κυρία Πρόεδρε, να πω ότι τα δύο επιπλέον κεφάλαια που πρόσθεσε ο εισηγητή νομίζω ότι είναι πολύ καλά, είναι πολύ καλέ οι προσθήκε αυτέ. Υπάρχει ένα κεφάλαιο για, τις, ε, ε, για τα θέματα μεταφοράς ενέργειας, για, τις, ε, για, τους πόρους. Θα κάνω και εγώ κάποιες προτάσεις, τους φυσικούς πόρους, θα κάνω και εγώ κάποιες προτάσεις ως προς αυτό. Πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε να βοηθήσουμε με τα υλικά ας πούμε, ας πούμε δάση και δασική πόρη, πώς τους χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Είναι μια εναλλακτική στα ορυκτά καύσιμα, για παράδειγμα. Ε, στο πέτρα-ελαιό κτλ. Είναι μια πολύ καλή εναλλακτική λοιπόν. Και θα ήταν ίσως καλός, ε, ένας ε, πολύ καλός τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους αυτούς με καλύτερο τρόπο. Έτσι ώστε να κάνουμε και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ήπειρος να, να συμβάλλουμε σημαντικά. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή για τις προτάσεις του και βεβαίως ευχαρίστω θα συνεργαστώ μαζί του για να εμπλουτίσουμε κι άλλο την έκθεσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Σιμάνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πριν ασχοληθούμε με τα ζωτικά θέματα της επανεκβιομηχάνησης, νομίζω ότι καλό θα ήταν να εξετάσουμε προσεκτικά τα αίτια των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Το μέλος της βιομηχανίας στην Ευρώπη μοιάζει αμφίβολο. Η βιομηχανική μας δραστηριότητα έχει συρρυκνωθεί. Τι συνέβη λοιπόν. Πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Γιατί έχει συνέπειες οικονομικής και κοινωνικής φύσης. Δεν νομίζω ότι το σχέδιο έκθεσης ε, απαντά σε αυτήν την ερώτηση ολοκληρωμένα ακόμη. Γίνεται λόγος για νέους κανονισμούς, προσδοκίες, ε, νέα προνομιακή μεταχείριση για τον έναν ή τον άλλον βιομηχανικό τομέα, όμως δεν δίδεται πραγματικά απάντηση στο ερώτημα για το τι συνέβη στη βιομηχανία μας. Ε, μόνο ο ακαδημαϊκός κόσμος μπορεί να μας δώσει ίσως μια απάντηση. Συχνά λέγεται ότι ε, μια από τις αιτίες είναι το υψηλό εργασιακό κόστος. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αλλάξουμε στην Ευρώπη, δεν εξαρτάται μόνο από μας. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας πέφτει λόγω και των υψηλών τιμών ενέργειας. Εδώ όμως μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές. Επίσης υπάρχει υπερβολική ρύθμιση. Η βιομηχανία στην Ευρώπη δυσκολεύεται πάρα πολύ. Μόνο όταν βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα θα αρχίσουν να εισραίουν περισσότερα χρήματα. Και μόνο τότε θα μπορέσουμε να σκεφτόμαστε να δαπανίσουμε το 3% του ΑΕΠ στην καινοτομία. Διαφορετικά ε, τα δημόσια οικονομικά μας δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πρόκληση οι μικρές επιχειρήσεις, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τότε μόνο θα μπορέσουν να έχουν χρήματα διαθέσιμα για να τα επενδύσουν στην έρευνα και την τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτό είναι προϋπόθεση για την επιτυχία. Ίσως να υπάρχουν πολλές καλές λύσεις για την πράσινη ενέργεια και τις πράσινες λύσεις, αλλά χρειάζονται χρήματα και αυτή τη στιγμή δεν τα έχουμε αυτά τα χρήματα γιατί δεν είμαστε παρκώς ανταγωνιστικοί. Ε, και υπάρχει και ένα τέταρτο αίτιο. Η έκθεση ε, ε, εστιάζεται στο πώς να εξοικονομούμε ενέργεια. Σωστό είναι αυτό. Αλλά και η πλευρά της προσφοράς είναι εξίσου σημαντική. Πώς θα παράξουμε φθηνή ενέργεια. Πώς θα διοχετεύσουμε φθηνότερες τιμές ενέργειας στην αγορά. Ε, εμείς έχουμε πολιτικές που συνεπάγονται υψηλές τιμές στην ενέργεια. Φοβάμαι ότι η λύση που έχουμε σήμερα δεν είναι καλή, δεν αρκεί, δεν συνάδει με την κατάσταση που επικρατεί στη Νότιο Ευρώπη. Στις νότιες χώρες ε, τα δημόσια οικονομικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε δινή θέση. Πρώτα όμως θα πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της δύση και του κέντρου της Ευρώπης ε, σε σχέση με, τη, με το ενεργειακό δυναμικό μας. Γιατί το ενεργειακό δυναμικό μας είναι τεράστιο και νομίζω ότι αυτό δεν τονίζεται παρκώς στην έκθεση. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως είπαμε την υπερβολική ρύθμιση και τις υψηλές τιμές της ενέργειας, αλλά δεν χρησιμοποιούμε παρκώς τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να απαντήσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν, το, αν καταφέρουμε να δώσουμε απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, η πράσινη βιομηχανία και η πράσινη... Ο λόγος στον κύριο Λάγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση του κυρίου Μπιούτι Κόφερ πραγματικά είναι εξαιρετική γιατί κάνει δύο πράγματα. Από τη μία τονίζει ότι μιλούμε για ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική και έτσι μιλά για ολοκλήρωση μεταξύ ευρωπαϊκού και κρατικού ε, επίπεδου. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό και απαραίτητο γιατί κατά τα λοιπά δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα να έχουμε μια ολοκληρωμένη ενιαία πολιτική. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό και σαφές ότι η εκβιομηχάνηση στα διάφορα κράτη-μέλη είναι τελείως διαφορετική, εξελίσσεται πολύ διαφορετικά και μπορούμε να την ελέγξουμε μόνο αν την δούμε από κοινού. Το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο της έκθεσης του κυρίου Μπουτικόφερ είναι ότι επικεντρώνεται σε πολύ κεντρικού τομεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχει νόημα να ε, κάνουμε ένα, μια πολύ ωραία ανθοδέσμη με διάφορα μέτρα, απαιτήσει, ευχές κτλ. Και να αφήσουμε τα σημαντικά στην άκρη. Οπότε εγώ υποστηρίζω απόλυτα τον κύριο Μπουτικόφερο όταν λέει ότι ένας από τους βασικούς ε, ογκόληθους που πρέπει να ε, τονίσουμε είναι αυτή η επιθετική πολιτική που πρέπει να, η προθετική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί μιλούμε και για την ε, έλλειψη καινοτομία, η οποία επίσης αποδυναμώνει την εκβιομηχάνηση. Ε, μιλήσαμε για την ε, επιθετική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε και θα ήθελα εγώ να πω ότι στην έκθεση της Κομισιόν για την καινοτομία αναφέρεται ότι υπάρχουν διάφοροι δείκτη, δείκτες, έρευνες, κορδίλια, κλάστερς, καινοτομίες κλπ. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην πολιτική μεταξύ της, ε, εντός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ ψηλά στην πολιτική κοινοτομία και κάποια άλλα πολύ χαμηλά. Γι' αυτό ε, πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Μετά, εσωτερική αγορά. Ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, ας πούμε στον τομέα που αφορά την στρατηγική για το εμπόριο, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο οξύ στη διατύπωσή μας και στην Κομισιόν, στην, δυνατότητα, ε, στην απονομή των εντολών που θα δώσουμε για τις διαπραγματεύσεις, να, ζητήσουμε να είναι πιο επιθετική, πιο απαιτητική σε ό,τι αφορά τι ε, επενδύσεις, σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με άλλε διεθνεί επιχειρήσει. Βεβαίως θα πρέπει να ελέγξουμε και το τι γίνεται με το dumping και ευρωπαϊκών και άλλων επιχειρήσεων. Μετά το θέμα της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας των πόρων, της ενεργειακής απόδοσης, ε, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ε, ε, έχουμε στην, τα έχουμε στην, στο δικό μας τον, στη δική μας την ατζέντα. Μιλούμε για την μείωση κατά 20% στα σημεία 57-59 ε, θα μπορούσε ο κ. Μπουτικόφερ να τονίσει ότι η Κομισιόν πρέπει να λάβει πιο σοβαρά την ευθύνη της, γιατί θέλουμε ένα σταθερό πλαίσιο, εφαρμογή δηλαδή της οδηγίας για την ε, ενέργεια και τις κατευθυντήριες γραμμές, ανανέσιμες πηγές ενέργειας, δυνατότητες της αγοράς. Αν η Κομισιόν λοιπόν έχει την ευθύνη, για την εκβιομηχάνηση θα πρέπει να λάβει και τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι αφορά την, απόδοση, την ενεργειακή απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μενίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω επιτέλους. Επιτέλους μιλάμε για την νέα εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Συζητάμε ένα κρίσιμο ζήτημα για τις χώρες μας και για την Ήπειρό μας. Παρ' όλα αυτά, αν δούμε λίγο αναδρομικά τι έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν θα πρέπει ούτε να μας καθησυχάζει, ούτε να μας κάνει ιδιαίτερα αξιόπιστους ε, οι πολιτικές μας ε, είμαστε για την εκμηχάνηση είναι ε, της δεκαετίας του 70. Τότε λέγαμε ότι μόνο μια ανταγωνιστική βιομηχανία θα μπορέσει να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την ή της ε, θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ακολούθησαν πάρα πολλές λευκές βίβλοι, το 80, το 90, το 2000, το 2010 και δεν είναι πλήρης ο κατάλογος. Έχουμε πάρα πολλούς ε, πηχαίους τίτλους για να μιλήσουμε για νέα προσανατολισμό της βιομηχανίας μας. Πρέπει όμως να κάνουμε την εξής διαπίστωση. Ο παραγωγικός μας ε, ιστός εξακολουθεί να μειώνεται και δεν έχουμε τα μέγιστα δυνατά εισοδήματα. Έκλεισαν εργοστάσια, ε, και ε, ξεχάσαμε και την έννοια του συλλογικού συμφέροντος. Οι χώρες μας σε διεθνές επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους ενώπιον των υπολείπων και εξακολουθούν να γίνονται μετεγκαταστάσεις. Για το λοιπόν θα πανούμε τόση ενέργεια και τόση σκέψη για να μην μπορούμε να καταφέρουμε να βγει από αυτό το ε, τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Όλοι οι προσανατολισμοί, όλα όσα κάναμε μέχρι τώρα ε, ήταν ε, σε μία, ένα πλαίσιο φιλελεύθερης συνένεσης. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε θέληση, δεν καταφέραμε να σκεφτούμε τι θέλει το συλλογικό συμφέρον για τη βιομηχανία και να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στις αγορές αυτού του μηχανισμού. Στα πλαίσια των ετών άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν οι όροι, αλλά η λογική που επιβάλλει ότι η αγορά είναι αυτή που καθορίζει ποιο θα επιβιώσει και ποιο θα πεθάνει είναι η ίδια. Ήρθαν πάμπολοι επιτροποί εδώ στην Επιτροπή μα να μα πούν τα ίδια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία ε, περιμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Ήγηκε η ώρα λοιπόν να αλλάξουμε λογική και να αλλάξουμε τη σημερινή συζήτηση, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μία ακόμα χαμένη ευκαιρία. Θα πρέπει να δώσουμε μια λύση στους λαούς μας. Αυτό χρειαζόμαστε και από κοινωνικής και από οικολογικής σκοπιάς, να αναπτύξουμε τη βιομηχανία, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές, οι οποίες υπάρχουν ήδη και να τις εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει dumping, πρέπει να σταματήσει το dumping και να μην ε, ε, ξεχνούμε ότι πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ε, σχεδιασμός ε, και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να συνεισφέρουν και αυτοί διότι έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρία να το κάνουν. Η βιομηχανία έχει ένα μέλλον στην Ευρώπη αλλά για να είναι πραγματικό δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε απλώς στα χέρια των μετόχων ε, και στα συνταξιοδοτικό ταμεία που θεωρούν όλα ότι πρέπει να προσμετράνται σε ποσά και σε απολύσεις για να μπορούν να επιτύχουν το στόχο τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να πω ότι χαίρομαι πολύ που ο εισηγητής ε, επικεντρώνεται στη βιομηχανική πολιτική. Εμείς υποστηρίζουμε όλα τα μέτρα που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας για την εσωτερική αγορά, τη γνώση, την έρευνα, την καινοτομία, την χρηματοδότηση κλπ. Επίσης, είναι σημαντικό στους τομείς που θα εργαστούμε να επικεντρωθούμε στις ε, αποδοτικές ε, πολιτικές που έχουμε. Ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Από τη μία έχουμε την πολιτική βούληση, από την άλλη έχουμε την πραγματικότητα, τη βιομηχανία. Όλοι θέλουμε καλύτερα πρότυπα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά τα καλύτερα πρότυπα, τα πιο υψηλά πρότυπα δεν σημαίνουν κατά ανάγκη και περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας μόνο μέσω αυτών των προτύπων. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτά τα μέτρα που όντως δημιουργούν και θέσεις εργασίας. Πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Γιατί η πολιτική, τα πολιτικά ευχολόγια δεν είναι επαρκή και δεν θα μας οδηγήσουν εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Η πολιτική μας πρέπει να είναι σαφής, απλή, στόχοθετημένη και στέρεα. Επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε διοικητικά ζητήματα και όχι στην επίτευξη των στόχων μας. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι η βιομηχανία μας συνδέεται με το παγκόσμιο περιβάλλον. Δεν είμαστε ε, μια αυτάρκης οντότητα εδώ στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι γίνεται, στα κοινωνικά και στα, ε, τι γίνεται με τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα αλλού, εκτός Ευρώπης. Γιατί τα πολύ μεγάλα κενά μπορεί να οδηγήσουν σε ε, χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλή βιομηχανική διπλωματία, καλές σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις εμπορικές μας σχέσεις, ε, την, ε, τις πρότασίλες την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας και επίσης να πω ότι στην Ευρώπη θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μία βιομηχανία ε, εχμής. Θα πρέπει να διαφοροποιηθούμε από τους υπόλοιπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε και ανάπτυξη και ανεξαρτησία. Ρόιλ, Ευχαριστώ συνάδελφος Ρόιλ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση. Αξίζει τον κόπο να τη συζητήσουμε και εγώ υποστηρίζω και τη στοχοθέτηση που αναφέρεται για την ευρωπαϊκή πολιτική που πρέπει να ανακαλύψει και πάλι από την αρχή τη βιομηχανία. Γιατί εκεί υπάρχει πραγματικά τεράστια ανάγκη. Ε, στην... Ε, το έχουμε αφήσει πολύ να στα, στις καλέντες το θέμα αυτό. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το θέμα της καινοτομίας και της εσωτερικής αγοράς πρέπει να μπει στο πυρήνα της συζήτησης. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, συμφωνώ απολύτως, γιατί ακριβώς έτσι θα, βελτιωθεί στο μέλλον η βιομηχανία. Κρίμα, που, το κρίμα είναι ότι το μέλλον είναι όντως η καινοτομία, αλλά δεν ρίχνουμε κανένα, καμιά ματιά στο παρελθόν, για το γιατί δημιουργήθηκαν τελικά τόσα προβλήματα, γιατί η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετώπισε τόσα προβλήματα. Εμείς ε, οι πολιτικοί τα τελευταία χρόνια ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με το να μην δραστηριοποιούμεθα θετικά και να μην αφήνουμε την ε, βιομηχανία στην ησυχία της, αλλά να κάνοντας ακριβώς το αντίθετο, ε, με πολλές ρυθμίσεις, με πολλές διατάξεις, προσπαθήσαμε να την φρενάρουμε τη βιομηχανία. Και νομίζω ότι ε, αυτό θα πρέπει να το πούμε στην έκθεση. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι με τόσο, πολύ, τόσο πολλές λεπτομερείς ρυθμίσεις, διατάξεις, κανόνες. Εντάξει, κανόνες θα υπάρχουν πάντα, αλλά σε ποιο βαθμό θέλουμε να επιβαρύνουμε κι άλλο τη βιομηχανία. Ή μήπω πρέπει να μπούμε πια στην φάση όπου στην Ευρώπη θα λέμε θέλουμε να αφήσουμε την ε, βιομηχανία να αναπτυχθεί, να αναπνεύσει, να καινοτομήσει. Και σε πολλά σημεία λέγεται ότι η ανάπτυξη της ε, ε, βιομηχανίας είναι η πράσινη. Ε, αυτό πώς το λέμε, πώς μπορούμε να λέμε τι είναι καλό και τι όχι. Εμείς απλώς λέμε τι είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι θετικό και σε ποιο βαθμό πρέπει να, σε ποιο μέτρο πρέπει να αναπτυχθεί η βιομηχανία. Αλλά έτσι δημιουργείται, δημιουργούμε, έτσι όπως αναφέρεται στην ε, έκθεση, σε ε, νέες διατάξεις. Θέλω λοιπόν ε, να το, να το κάνουμε από την άλλη μεριά, να το κάνουμε αντίθετα. Να μην μιλούμε δηλαδή για μονομερείς διαπιστώσεις, δεν μιλούμε για την μελλοντική βιομηχανία μόνο. Ναι, είναι και αυτό σημαντικό. Αλλά εδώ θέλουμε να δούμε η βιομηχανία που έχουμε σήμερα πώς θα παραμείνει και πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω. Και αυτό νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας συνδέεται σε εισαγωγικά με την παλιά βιομηχανία, η οποία επίσης απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Να την αφήσουμε ξαφνικά και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με κάτι ε, καινούριο τελείω, νομίζω ότι είναι λάθος. Πρέπει τις, ε, τις δυνατότητες που έχουμε να τις ενισχύσουμε πολύ περισσότερο και βεβαίω από τις δυνάμει μας και από τα ατού μας να δημιουργήσουμε και κάτι νέο. Αλλά το θέμα δεν είναι να έχουμε μεμονω... επιμέρους ή μεμονωμένες ε, διαπιστώσεις. Ε, αυτό είναι μόνο το σημείο κριτικής που θα ήθελα να αναφέρω. Ε, η στοχοθέτηση ναι, στη βιομηχανία σωστή, στοχοθέτηση για τη βιομηχανία που θέλουμε να πάμε, σωστό και για την εσωτερική αγορά και για την καινοτομία, ναι, αλλά για τα υπόλοιπα σημεία θα ήθελα να γίνουν κάποιες διορθώσεις, τις οποίες θα υποβάλω με κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Τζέρεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όταν μιλούμε για βιομηχανία, μιλούμε για υλική παραγωγή. Παραγωγή εμπορευμάτων. Στον τομέα αυτό πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πυροδοτούν την ανταγωνιστικότητα. Το κόστος της ενέργειας, το κόστος των πρώτων υλών και η κατάσταση επίσης εξαρτάται από, από την οργάνωση του εργατικού δυναμικού. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες της ανταγωνιστικότητας. Εάν δούμε την ανταγωνιστικότητα σφαιρικά, θα καταλάβουμε ότι η Ευρώπη υπολείπεται από τις άλλες χώρες. Είναι πολύ λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τους εταίρους της. Η ενέργειά μας ε, έχει διπλάσεις και τριπλάσεις τιμές σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, όσο αφορά τις πρώτες ύλες, είτε δεν έχουμε επειδή τις έχουμε υπερεκμεταλλευτεί, είτε είναι πολύ ακριβές. Και με την εξαίρεση της Γερμανίας η οργάνωση του εργατικού δυναμικού ε, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Τι, να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε για να υπερκεράσει τα εμπόδια η βιομηχανία. Καταρχήν να δούμε το θέμα της μετεγκατάστασης της παραγωγικής δυναμικότητας. Δεύτερον, έχουμε πολυεθνικές, έχουμε μεγάλους ομίλους οι οποίοι ε, προς, καταφεύγουν σε φορολογικούς παραδο, παραδείσους και συχνά η, παράδειση, φορολογική παράδειση αυτή επιβάλλουν τους δικούς τους όρους. Ε, η βιομηχανία τους επιλέγει βέβαια επειδή τη βολεύουν. Στη συνέχεια έχουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται τοπικά. Ε, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν καλύτερα εάν δραστηριοποιούνταν μέσα σε μια καλύτερη ατμόσφαιρα, εάν μπορούσαν να απασχολούν ε, τοπικούς ανθρώπους, αν μπορούσαν να βρουν πρώτες ύλες ε, από κοντινές αποστάσεις και αν την χέναν της κατάλληλης ε, στήριξης από τις περιφέρειες. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, μπορούμε να, κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, να το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο και να οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσπαθήσουν ε, να αναπτυχθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο των εθνικών τους συνόρων. Αλλά πολύ σωστά ο εισηγητής τονίζει ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτημα όμως είναι πώς. Πώς θα διαμορφώσουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα εδώ. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία γιατί αν δεν το κάνουμε τότε θα συρρυκνωθεί και θα εξαφανιστεί τελείως δεν, αν δεν έχουν τη βάση, αν δεν έχουν τους εργαζόμενους που χρειάζονται οι βιομηχανίες, ε, εάν πρέπει να πάνε σε άλλες χώρες για να βρουν μια καλύτερη δασμολογική, φορολογική πολιτική. Πώς θα τη συγκρατήσουμε εδώ τη βιομηχανία. Ξέρουμε ότι είμαστε ευάλωτοι και ταυτόχρονα μας περιφρονούν. Πρόκειται για ένα οξύμορο σε αυτό το τομέα, αυτή η καινούργια εκβιομηχάνηση της Ευρώπης πρέπει να είναι περιφερειακή, να χρησιμοποιεί περιφερειακούς εργαζόμενους και περιφερειακή. Ευχαριστώ κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να συγχαρώ τον κύριο Μπουτικόφερ, ο οποίος ε, αντιμετώπισε πάρα πολύ εύστοχα ένα τόσο σημαντικό ζήτημα εν καιρό κρίσης θεωρώ ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε και τον συνάδελφο Λάγκε, ο οποίος ε, ασχολήθηκε και αυτός με το ζήτημα. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στην καινοτομία, αναφερόμαστε και ε, στην ανάγκη ανάπτυξης ε, της καινοτομίας. Και νομίζω ότι δίνεται ιδιαίτερη ένταση τις ε, ενεργείες εχμέης και στα καινοτόμα προϊόντα. Δεν ε, μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι χωρίς βιομηχανία θα λειτουργήσει καινοτομία. Στο βιομηχανικό κόσμο Φαίνεται όμως ότι δεν έχει παρισφρήσει η διαδικασία της καινοτομίας πολλές φορές αναφερόμαστε στα κατάλληλα επιχειρηματικά μοντέλα. Το θέμα όμως είναι πώς ε, θα ε, τοποθετηθεί στην αγορά ένα νέο προϊόν. Και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την καινοτομία του προϊόντος. Μια βιομηχανία που παράγει ένα κακό προϊόν ε, σίγουρα δεν έχει μέλλον. Πρέπει λοιπόν να δούμε το κατάλληλο επιχειρηματικό, το κατάλληλο εμπορικό μοντέλο και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο καλύτερα πώς θα παρουσιάζονται στην αγορά νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα. Ε, όλο ένα και περισσότερο σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια τάση στη στρατηγική Ευρώπη 2020 να ε, δίνουμε έμφαση στην πτυχή της τεχνολογίας, την οποία χρειαζόμαστε μεν, αλλά αυτή θα πρέπει να συνάδει και να συμβαδίζει με νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και διάφορα άλλα μοντέλα τα οποία ναι μεν... Ε, δεν είναι τόσο προχωρημένα, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και άλλες δυνατότητες σε φορολογικό επίπεδο, να άρουμε κάποιους φραγμούς, ε, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα στην εσωτερική αγορά. Ε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εξακολουθούν να επιμένουν, ε, δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό, θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται στους εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού και να επιμείνουμε και στην ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει να ευνοούνται οι θέσεις εργασίας ε, και να ε, δίνει νέα όθηση στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε τα ζητήματα. Ε, υπάρχει μια περιφερειακή πολιτική η οποία θα πρέπει να ενταχθεί και στα πλαίσια των φιλοδοξιών που μας παρουσίασαν οι βιομηχανίες μας. Τίθεται και θέμα επενδύσεων βεβαίως. Αναφερόμαστε συνεχώς σε επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά προς την κατεύθυνση της καινοτομίας μεν, αλλά γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και το ρόλο που διαδραματίζουν όλες οι επιχειρήσεις, και οι μεγάλες και οι μικρές. Και επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο Νότο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού ιστού και αυτό θα πρέπει να το διατηρήσουμε και στο Νότο ε, και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και στις νότιες περιοχές πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτά σας ευχαριστώ για την έκθεση κύριε Μπουτικόφερ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπουτικόφερ Εγώ αντιλαμβάνομαι με το δικό μου προσωπικό τρόπο την παρούσα κατάσταση. Επιτέλους έχουμε μια βιομηχανική πολιτική, διότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι η ε, παραγωγή ήταν κάτι ξεπερασμένο και το μέλλον ήταν στην οικονομία. Είδαμε τι προκάλεσε αυτό και διαπιστώσαμε επίσης ότι σε τομείς στους οποίους δεν συνέβη αυτό, όπως για παράδειγμα στον αεροδιαστημικό τομέα, υπάρχει ανταγωνιστική ε, βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευπρόσδεκτη λοιπόν επιτέλους η επιστροφή της βιομηχανικής πολιτικής. η οποία θα μας δώσει και μια κατάλληλη πορεία ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και την ε, βιομηχανική μας ε, νοοτροπία αλλά και την ανταγωνιστικότητα γιατί και στην Κίνα θα υπάρξει αύξηση του κόστους εργασίας και επομένως εμείς πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάλειμμα των 10-15 ετών χωρίς ταυτόχρονα να χάσουμε και την ε, ε πτυχή που έχουμε της βιοτεχνίας. Παραδείγματο χάρη, στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάνελ έχουμε ανταγωνισμό με την Κίνα γιατί πουλά κάτω του κόστου ε, σε σχέση και με την ίδια του την παραγωγή. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το εξετάσουμε γιατί μπορεί αυτό να σημαίνει και ότι η Κίνα θα θέλει να γίνει ο κατασκευαστής του κόσμου. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε διότι δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από άλλους για τομείς οι οποίοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Υπάρχει και ένας επαναπατρισμός της βιομηχανίας. Αυτό το διαπιστώνουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε και θα πρέπει λοιπόν και εμείς να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική η οποία αφενός σημαίνει ότι θα πρέπει η φορολογία να πεάει από την εργασία στην κατανάλωση των πόρων, επομένως δεν θα πρέπει να απαραίτητος οικολογική οικονομία, αλλά θα πρέπει να είναι αποτελεσματική όσον αφορά τους πόρους και την εργασία. Αυτό άλλωστε θα εξετάσουμε και στο επόμενο σημείο όταν θα μιλήσουμε για την ε, ε, άμυνα και την βασική, τη βιομηχανική βάση της ευρωπαϊκής άμυνας. Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη βιομηχανική πολιτική και να υπάρχει ευρωπαϊκή διάσταση την οποία υπενθύμησα για την ε, αεροδιαστημική βιομηχανία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κοφεύουμε και να μιλήσουμε επιτέλους για την βιομηχανική πολιτική. Η κυρία Μαζεκούκοτς. Να ευχαριστήσω και εγώ τον εισηγητή. Το βασικό ερώτημα που έχω για τούτη την ε, έκθεση είναι πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτά τα ε, προϊόντα από τη δική μας την αγορά των 500 εκατομμυρίων σε μια αγορά 7 δισεκατομμυρίων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό και πού βρίσκεται η κατάσταση. Η βιομηχανία αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια και δεν έχει πάρα πολλά κίνητρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τους τομείς που είναι ελκυστικοί. Δεν θα πρέπει να πούμε εμείς, να υποδείξουμε στη βιομηχανία τι να κάνει ας πούμε, η ε, φαρμακολογία, η, ε, η, ενεργεια, πληροφορία σε σχέση με την, ε, με την ενέργεια. Όλα αυτά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να δούμε πώς έχουν τα πράγματα ανατομέα στην Ευρώπη, αν θέλουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτή την αγορά των 7 δισεκατομμυρίων ατόμων. Πρέπει να μειώσουμε τον ανταγωνισμό μεταξύ μας και να προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όταν μιλούμε ε, για τη θέση μας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί λοιπόν, ε, ε, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κέντρα αριστείας μας για να μπορέσουμε να εισχωρήσουμε στην παγκόσμια αγορά και στο Connecting Europe έχουμε μια μελλοντική ε, χρηματοδοτική προοπτική που θα είναι ιδιαίτερο υποφελής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα σύνδεση εσωτερικά, για να μην μιλήσω για την εξωτερική τους σύνδεση. Οπότε πρέπει να ε, θέσουμε σωστές προτεραιότητες. Δεν έχουμε αρκετούς μηχανικούς, δεν έχουμε αρκετούς εμπειρογνώμονες. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε εμείς το δικό μας εμπορικό σήμα, το Made in Europe. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω τη δουλειά του συναδέλφου Μπίτικόφε και την παρέμβαση του φίλου Φρανκ Προύστ που προέρχεται που έχει διπλή ιδιότητα ε, και θέλω να μείνω εδώ γιατί ε, στην Ευρώπη ε, εκπροσωπείται το 8% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 23% του οικονομικού ε, πλούτου και το 70% των δημόσιων οικονομικών. Στις συνθήκες αυτές πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να περιλάβουμε το σύνολο των δημόσιων οικονομικών μας. Άκουσα αυτά που είπε ο, εξ, που είπε ο εξαιρετικός συνάδελφος. Άλλοι βλέπουν την αγορά ως πρόβλημα. Εμείς βλέπουμε την αγορά ως λύση. Αλλά υπάρχει μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Κάθε φορά που οι σοσιαλιστές, Πασκαλαμή και λοιποί, στα κράτη-μέλη είναι σοσιαλιστές, ε, όταν όμως συμμετέχουν στα υπερεθνικά όργανα γίνονται σούπερ φιλελεύθεροι. Και μιλούν πάντοτε για διοικούμενη οικονομία, διαχειριζόμενη οικονομία. Αλλά ο πολίτης τι βλέπει. Βλέπει την οικονομία των βιομηχανιών. δεν είναι μόνο ότι το λέμε στη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στηριχθεί πάρα πολύ στην κατανάλωση. Εγώ χαίρομαι που τώρα επιτέλους ενδιαφέρεται για την παραγωγή βιομηχανική, γεωργική. Ε, ανήκω σε μια εκλογική περιφέρεια όπου ακόμα τελούμε υπό το σοκ της άρνησης ε, της ε, ε, Ευρωπαϊκής Κομισιόν να συμφωνήσει στην συγχώνευση δύο μεγάλων βιομηχανικών κολοσσών. Αν θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές στον κόσμο και με υπεργολαβίες και με τα λοιπά, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτού του τύπου οι αποφάσεις είναι που δεν τις ανέχεται πια ο Ευρωπαίος πολίτης. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι οι βιομήχανοι όταν μας ακούν έχουν πια βαρεθεί την ε, πολιτική αστάθεια. Ε, υπάρχουν κανόνες, αλλά κάθε τρεις και πέντε τους αλλάζουμε για την υγεία, για το περιβάλλον, οι κοινωνικοί κανόνες. Χρειάζονται όλα αυτά, αλλά χρειάζεται και σταθερότητα. Τέλος, να θέσω στην προσοχή του εισηγητή το θέμα του νομίσματος. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχει ο πόλεμος των νομισμάτων. Πρέπει η διαχείριση του νομίσματός μας, λοιπόν, να εξυπηρετεί το συμφέρον της βιομηχανικής πολιτικής. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ ισχυρό το ευρώ. Ε, ξέρω ότι είμαι αρκετά απομονωμένο πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό που μας λένε όμως οι βιομήχανοι τι είναι. Προσοχή στην νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική κύριε Τρισέ με όλες αυτές τις κρίσεις 2008-2009 υπάρχουν ανεξάρτητες ε, μελέτες που λένε 0% ε, ανάπτυξη με διπλάσια επιτόκια από αυτά που βλέπουμε στην Αμερική. Με συγχωρείτε ξέχασα για το παγκόσμιο εμπόριο. Να μην είμαστε πια να προσέξουμε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο εμπόριο. Εκεί θα, από εκεί θα προκύψουν οι λύσεις. Ευχαριστώ, Κρίστιαν Χέλλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήδη υπόθηκαν πολλά. Ένα γενικό σχόλιο θέλω να κάνω για κάποια επιμέρους σημεία. Είμαι αρκετά προσεκτικός για το θέμα της ε, ε, βιομηχανικής πολιτικής. Τη βιομηχανική πολιτική ε, ούτε στην Ασία, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ευρώπη στο παρελθόν την είδαμε να είναι πολύ επιτυχής. Υπήρχαν κάποια πράγματα όπως η φορολογία ας πούμε, που δεν ήταν πολύ, πολύ επιτυχής. Αν δούμε εκθέσεις του ε, όσα ε, φαίνονται τα στοιχεία. Έχουμε πάρα πολύ μικρές επενδύσεις στον τομέα, έχουμε ε, επίσης μειούμενη εκπαίδευση για τον τομέα, ετοιμότητα σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ετοιμότητα ως προς τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία επίσης πολύ μικρή. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τομείς πολύ βασικοί. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να τους συνδυάσουμε με την βιομηχανική πολιτική ή αν θα πρέπει να τους δούμε μεμονωμένα. Για αυτά τα σημεία λοιπόν, μάλλον θα πρέπει κάπως να αλλάξουμε τα πράγματα. Οι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί με να είναι περιορισμένε, αλλά θα πρέπει στην έκθεση να είναι πολύ συγκεκριμένο το τι θέλουμε να κάνουμε. Μιλούμε για τον ορίζοντα 2020 ε, που θα είναι το πρώτο πρόγραμμα όπου δεν θα αυξηθεί ποσοστιαία η ε, έρευνα, αλλά μάλλον θα παγώσει στα τωρινά νούμερα. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το κοινοβούλιο που έχει ένα πολύ γνωστό ρεκόρ στο πόσο ρυθμίζει μπορεί να διορθώσει το ζήτημα αυτό. Θέλουμε να μειώσουμε την ρύθμιση, της ε, κατευθυντήριας γραμμές. Σε πολλούς ε, τομείς πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας. Και κάνουμε πολλές φορές συζητήσεις πολύ βασικές. Ας πούμε δεν συμφωνούμε να δούμε την ε, βιομηχανία ως, ως μεγάλη βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως δύο χωριστά πράγματα δηλαδή. Μιλούμε ε, για μικρές επιχειρήσεις ε, συνήθως, δεν μιλούμε για μικρομεσαίες. Αλλά αν δείτε πού είναι η βιομηχανική παραγωγή ποσοστιαία, δεν βρίσκεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή, αλλά Επίσης δεν επηρεάζεται και πάρα πολύ και από, τις μεγάλες, από τους μεγάλους βιομηχανικούς κόλωσους που δραστηριοποιούνται παγκοσμίω. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε ποια είναι η βιομηχανία στην, στην Ευρώπη, αλλά εδώ εμείς στο Κοινοβούλιο δεν είμαστε στην, δεν, δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Μιλούμε πάντα για πολύ ε, ξεκάθαρα στατιστικά δεδομένα. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε εμείς να κάνουμε να μην μιλούμε μόνο έτσι, θεωρητικά, να δούμε και στην πράξη ποιε είναι οι δυνατότητε χειρισμού που έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Χίμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν στο θέμα της ανταγωνιστικότητας και πώς μπορεί να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα ε, αναφερθήκατε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση ως έχει. Θα πρέπει να εξετάσουμε ποιοι τομείς είναι δευτερεύοντες και ποιοι τομείς θα πρέπει να θεωρηθούν τομείς προτεραιότητας ίσως ε, σε κάποιους τομείς ε, να μην ε, πρέπει να συνεχιστεί η παραγωγή και να μπορούμε να κάνουμε απλώς εισαγωγή και να επικεντρωθούμε σε, τομείς, σε τομείς στους οποίους μπορούμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Δεν μπορεί να επιβαραβεύουμε συνεχώς τους εαυτούς μας, είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με αυτά που κάνουμε, ετοιμάζουμε συνεχώς νέα νομοθεσία η οποία στην πραγματικότητα καταρακώνει τη βιομηχανία. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε κάτι για το θέμα αυτό. Να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε πάντα φιλικά διακύμονοι προς την βιομηχανία. Τις περισσότερες φορές είμαστε εχθρικοί απέναντί της. Ε, τις περισσότερες φορές ετοιμάζουμε νομοθεσία η οποία βοηθά τη μετεγκατάσταση. Ναι, μεν ε, χαϊδεύουμε τα αυτιά της βιομηχανίας και της λέμε ότι θέλουμε να τη βοηθήσουμε, αλλά η βιομηχανία διαφεύγει σε άλλες χώρες παρόλα αυτά διότι δεν τη βοηθούμε. Και θα ήθελα να σταθώ και στο εξή. Υπάρχουν άλλες χώρες στις οποίες αναπτύσσεται η βιομηχανία και χάνουμε όχι μόνο τα εργοστάσια τα οποία κλείνουν, αλλά ε, στις περιοχές στις οποίες υπήρχαν παλιά εργοστάσια η γη αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε τρίτους. Νομίζω ότι θα πρέπει σαφώς να επισημάνουμε τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Υπάρχει και η σχετική διάσκεψη των μηχανικών που έγινε στην Πολωνία προσφάτως και ε, ήρθαν και κάποιοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αναφέρθηκαν στην ενέργεια η οποία θα παράγεται από μάχμα από το κέντρο της γης. Αυτά για μας είναι πυρηνική επιστήμη. Τι καθόμαστε λοιπόν και συζητάμε. Έχουμε μείνει πίσω... Ε, Αυτά γίνονται στις Ηνωμένε Πολιτείε και εμείς ε, δεν ξέρουμε τίποτα τι γίνεται. Χάνουμε την τεχνολογία μέσα από τα χέρια μας και πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να συγχαρεί τον εισηγητή, τον κύριο Μπουτικόφερ, διότι μας παρουσίασε κατά την άποψή μας μια πολύ ισορροπημένη και ενδιαφέρουσα έκθεση. Η έκθεση αντικατοπτρίζει πάρα πολύ καλά το πολύ καλό μήνυμα το οποίο θεωρούμε ότι διαβίβασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγινε ε, πολύ καλά αποδεκτό και από την κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βιομηχανία ήταν κάτι το οποίο είχε παραγωνιστεί στο παρελθόν και νομίζω ότι πλέον διαθέτουμε τα κατάλληλα στοιχεία για να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία της ε, ε, επανεκβιομηχάνησης της βιομηχανίας που είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να επιβιώσουμε εάν θέλουμε όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική στο μέλλον. Τρία στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Το πρώτο είναι η συνέπεια στη χάραξη της πολιτικής μας. Θεωρώ ότι η συνέπεια στη χάραξη της πολιτικής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ενισχύσουμε στο εγγύς μέλλον προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας. Και τι εννοώ. Εννοώ ότι θα πρέπει να υπάρχει οριζόντια ε, συνέπεια, καλύτερη συνέπεια μεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι κάτι το οποίο ο, δεν έλαβε τη δέουσα προσοχή στο μέλλον. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα, κάτι το οποίο χρησιμοποιείται και στην ε, ε, προετοιμασία κατά την ε, διαπραγμάτευση για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και από εκεί και πέρα υπάρχουν και αξιολογήσεις για το συλλογικό κόστος. Υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε. Το κόστος της ενέργειας. Πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να εξετάσουμε τις διάφορες συνιστώσεις. Ε, δεν είναι η μόνη συνιστόσα η ενέργεια, αλλά η συνιστόσα της ενέργειας ε, αλλάζει πλέον πορεία. Το κόστος της ενέργειας ε, παγκοσμίω δεν είναι υπέρ της βιομηχάνησης της Ευρώπης, επομένως θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να εμβαθύνουμε τη διαδικασία της αποτελεσματικότητας των πόρων στις κατασκευές και την ε, ε, ενεργειακή απόδοση και στη παραγωγή αλλά και για άλλους σκοπούς όπως για παράδειγμα την ε, ηλεκτροδότηση σπιτιών κτλ. Και τέλος κάτι το οποίο θα βρείτε στο τέλος της έκθεσης και θεωρώ ότι είναι υψής της σημασίας είναι το θέμα της σταθερής Ευρώπης κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε ποιες ήταν οι συνέπειες της κρίσης στην εσωτερική αγορά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Υπάρχουν πάρα πολλές ροχμές, τις οποίες έχουμε ήδη εντοπίσει. Είναι σαφής η κατάσταση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου οι ε, συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την εσωτερική αγορά και σε ποιο βαθμό οι ανισορροπίες ε, οι οποίες εντοπίστηκαν και οι οποίες σε κάποιο βαθμό ε, ήταν και στην πηγή του προβλήματος εξηγούν ή μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ ε, για να ξεκινήσει η οικονομική ανάκαμψη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουν δημιουργηθεί πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία προσφάτως τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ στην Ευρώπη χάνουμε θέσεις από αυτό το τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τα αίτια και θεωρώ ότι τα αίτια είναι βαθύτερα, γεγονός που σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλάβουμε περαιτέρω δράση κάποια στιγμή. Ε, προς το παρόν, να συγχαρώ και πάλι τον κύριο Μπουτικόφερ για την εξαιρετική του έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς, για να ολοκληρώσει τη συζήτηση, ο κύριος Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τα σχόλιά τους για τις παρατηρήσεις τους. Δεν είναι πολύ σημαντικό, σημαντική απλώ η συζήτηση που κάνουμε, αλλά είναι και πολύ θερμή. Ε, καταρχάς να πω, και αυτό είναι το πιο σημαντικό στη συζήτηση αυτή για μένα, ότι ευχαριστώ βεβαίως και όλους όσους το τόνισαν, ότι χρειαζόμαστε κοινό ευρωπαϊκό δρόμο. Όχι μόνο γιατί έχουμε την δυνατότητα ρύθμισης ή νομοθετησίας κτλ. Αλλά πρέπει να έχουμε μια κοινή κατανόηση, μια, ένα κοινό όραμα το οποίο πρέπει να προωθήσουμε. Γιατί αλλιώς όλα όσα κάνουμε σε μεμονωμένα, ε, μέρη, σε μεμονωμένα μέτρα θα παραμείνουν κενό γράμμα. Μιλήσαμε για συνοχή. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λέξη. Μιλήσαμε για οριζόντια πολιτική, αλλά και ε, συνδυασμό μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων. Γι' αυτό πρέπει να, έχουμε έναν, ε, να προχωρήσουμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δρόμο. Και αυτό το χρειαζόμαστε επίσης, γιατί ο κόσμος δεν μας περιμένει, δεν θα περιμένει μέχρι η Ευρώπη να λύσει τα δικά της, τα εσωτερικά της θέματα για να προχωρήσουν αν κοιτάξει κανείς την Κίνα ή τη ΣΥΠΑ ή την Κορέα ή την Ιαπωνία, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες σε ενεργειακό επίπεδο που γίνονται ώστε να εξυγχρονιστεί η βιομηχανία. Και αυτό δεν είναι απλώς προγράμματα πολύ μικρά ή ε, ίσονος σημασίας, είναι, είναι πολύ σημαντικά προγράμματα. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, γίνονται ε, πάρα πολλές ε, επενδύσεις ό,τι αφορά την κορεα η την ιαπωνια υπαρχουν παρα πολλες δραστηριοτητες σε ενεργειακο επιπεδο που γινονται ωστε να εξυγχρονιστει η βιομηχανια και αυτο δεν ειναι απλως προγραμματα πολυ μικρα η ίσονο σημασιας ειναι ειναι πολυ σημαντικα προγραμματα στην ιαπωνια ας πουμε γινονται παρα πολλες επενδυσεις οτι αφορα την ε, την, ε, τις επενδύσεις στην ενέργεια από εξόριξη. Ε, μιλάμε δηλαδή για την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, μέσω αυτού προσπαθούν να λύσουν το θέμα της ενέργειας. Εγώ είδα τα όσα είπατε, τα άκουσα πολύ προσεκτικά και πρέπει να πω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει η Ιαπωνία η Ιαπωνική βιομηχανία σε συνεργασία με την Ιαπωνική κυβέρνηση και πώς απαντά στις προκλήσεις. Θα πρέπει λοιπόν την εμπειρία βιομηχανικών ανταγωνιστών μας να τη χρησιμοποιήσουμε, όχι να την, όχι να την υπονομεύουμε. Δεν είναι σωστό να υπονομεύουμε τον αντίπαλο, μπορούμε να μάθουμε από αυτόν. Και επίσης, δεν θεωρώ ότι ο στόχος ε, που έχει βάλει η Κομισιόν έτσι γενικά στην ανακοίνωσή της έχει τύχει θετικής αντιμετώπισης. Το τι γίνεται δηλαδή με την αύξηση του, της βιομηχανικής παραγωγής σε σχέση με το ΑΕΠ για την αύξηση του 20%. Αυτό δεν θα γίνει μόνο με τα μέσα που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι. Και αυτό που δεν κατάλαβα και απλώς το αναφέρω σε κάποιους συναδέλφους, είπανε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον ανταγωνισμό, την ανταγωνιστικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θα πει αυτό. Θα πει ότι δεν θα πρέπει να εμβαθύνουμε την εσωτερική αγορά. Αν είναι αυτό το μήνυμα που θέλετε να στείλουμε, ε, εντάξει, είναι και αυτή μια εναλλακτική τώρα, για τα όσα είπαμε, για τα λάθη που έχουμε κάνει και τα λοιπά, το είπε και ο κύριος Ρόιλ. Ε, συμφωνώ, συμφωνώ, ε, είμαι ένοχος. Ε, δεν έκανα πολύ καλή κρίση, ανάλυση της κρίσης, πλήρη και περιστατωμένη, αλλά αυτό δεν μπορείτε να το περιμένετε και σε μια έκθεση με πολύ συγκεκριμένους χαρακτήρες. Οπότε, Τώρα δεν θα πρέπει να αρχίσουμε απλώς να ε, ψάχνουμε από εδώ και από εκεί. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τον ε, δείκτη καινοτομία του Bloomberg που μιλά για τις 10 ε, καλύτερες χώρες. Στις 10 top χώρες οι 6 είναι ευρωπαϊκές χώρες. Έξι ευρωπαϊκές χώρες λοιπόν βρίσκονται στο top 10 του Bloomberg για, τις, ε, για την κοινοτομία. Οπότε έχουμε πάρα πολλέ δυνάμεις πάνω στι οποίε μπορούμε να στηριχτούμε για να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι θα ήταν λάθο η ανάπτυξη που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ξαφνικά να, να, να την υποβαθμίσουμε. Πού είναι οι δυνάμεις μας, πού είναι τα ατού μας, ποια είναι τα, τα παραδείγματα που ήταν ε, επιτυχή. Η Δανία, η Σουηδία, η Αυστρία, η Φιλανδία, η Γερμανία. Είναι υποδείγματα που έχουν ε, αξιολογηθεί πάρα πολύ καλά σε αυτούς τους δείκτες. Και αυτοί επίσης ανήκουν στην ευρωπαϊκή ε, βιομηχανική πολιτική δεν θα πρέπει να μπούμε ο καθένας πίσω από, την, από το εθνικό του συμφέρον. Θα πρέπει να συνδυάσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις επιτυχίες μας, από όπου και αν προέρχονται. Ναι, πρόεδρε, χτυπάτε και το σφυράκι σας. εντάξει, να κλείσω. Θα σταματήσω εδώ. Οπότε ε, δεν απάντησα σε όλου ε, και ρίχνω την ευθύνη σε εσά γιατί εσεί με σταματήσατε, κυρία Πρόεδρε. Οπότε α μην με κατηγορήσουν οι συνάδελφοι. Ε, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους για τι απαντήσεις που δεν πρόλαβε να δώσει ο κύριος Μπιουτικόφερ. Μέχρι τις 19 Ιουλίου στις 12 η ώρα είναι η προθεσμία για την υποβολή πρωτοπολογιών. Και τώρα ο κύριος Μπιντι πάνω στο σχέδιο του προϋπολογισμού 2014. Θέμα που πρέπει να λύσουμε μέσα σε λίγα λεπτά νομίζω. Okay, me again, colleagues. Um, this is about the, um, Εγώ και πάλι συνάδελφοι. Πρόκειται για τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο προπολογισμού τον Ιούνιο στις 26 Ιουνίου. Τα προτινόμενα επίπεδα δαπανών ε, αντανακλούν ε, τα ανώφλια, το, το, τα ανώτατα όρια, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη το Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Σε γενικές γραμμές αυτός ο νέος προϋπολογισμός για το επόμενο έτος επιφέρει μία ετήσια μείωση των κονδυλίων της σε όλα τα κεφάλαια σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013 με εξαίρεση το 1α, το κεφάλαιο, τον τίτλο 1α. Αλλά έχει σημασία να σημειώσουμε ότι η αύξηση που βλέπουμε στο 1α απορροφάται από τα μεγάλα έργα υποδομών και από το χρηματοδοτικό μέσο διασυνδέοντας την Ευρώπη. Ε, τα υπόλοιπα υποκεφάλαια, με εξαίρεση τα τρία κύρια έργα υποδομών, μειώνονται ε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε ετήσια βάση. Αν μπορώ να επαναλάβω κάποια πράγματα που είπαν συνάδελφοι στην προηγούμενη συζήτηση για την σημασία της ανάπτυξης και της καινοτομίας, αυτός ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος ε, ε, δεν βάζει τα χρήματα στο σωστό μέρος η Επιτροπή έχει θέσει κάποια πολιτική έμφαση για την ανεργία των, στην ανεργία των νέων και μέτρα καταπολέμησής της με τις εμπροσθοβαρείς ε, προσεγγίσεις, ε, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και εκεί κάποιες εμπροσθοβαρείς κινήσεις προτείνονται. Ο προϋπολογισμός είναι λίγο περίπλοκος δεν αντιστοιχούν όλες, όλοι οι, τίτ, οι ειδικότεροι τίτλοι, τους ειδικότερους τίτλους των προηγούμενων προϋπολογισμών και δεν έχουν λυθεί και όλες ε, οι λεπτομέρειες σχετικά με τα καινούργια κονδύλια. Χρειάζονται κάποιες πρόσθετες διευκρινήσεις και νομίζω πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει αυτές τις διευκρινήσεις να μας ε, δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όσο το δυνατόν συντομότερο. Όσο το δυνατόν συντομότερα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, με βάση τους αριθμούς που έχουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε να καθορίσουμε πόσα χρήματα θα, θα διοχετευθούν στις πρωτοβουλίες GDI το 2014 από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Τώρα, πληρωμές. Οι πληρωμές των τελευταίων δύο ετών δεν έχουν <laughs> φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο όπως όλοι γνωρίζουν. Και αυτό θέτει σε κίνδυνο την υγιή δημοσιονομική διαχείριση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Χρειάζονται πρόσθετες πρέπει να επιτραπούν πρόσθετες πληρωμές για το 2013. Επίσης, το επίπεδο των πληρωμών για το 2014 επανέρχεται στο επίπεδο του 2012. Πράγμα που οφείλεται βέβαια στις ανάγκες που έχουμε και επιβάλλει μια αναθεώρηση. Κάποιες προτάσεις. Πρώτον, Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει περαιτέρω περικοπές και δεν το ξέρουμε ακόμη, γιατί το Κορεπέρ θα αποφασίσει μέσω της έγγραφης διαδικασίας στις 18 Ιουλίου και η ψηφοφορία στο Συμβούλιο θα γίνει στο ΕΚΟΦΗΝ στις 25 Ιουλίου. Εάν όμως το Συμβούλιο προτείνει περισσότερες περικοπές, προτείνω να αποκαταστήσουμε την πρόταση της Κομισιόν τουλάχιστον για τα κονδύλια 1α ε, που άπτονται των δικών μας αρμοδιοτήτων. Δεύτερον, προτείνω να αυξηθεί η εμπροστοβαρή κίνηση για το, οράζιον για το ορίζοντας 2020. Εάν γίνει τέτοια εμπροσ... υπάρχουν κάποιες εμπροστοβαρείς προσεγγίσεις, αλλά δεν αρκούν για να μειωθεί το χάσμα το, μεταξύ των προηγούμενων αριθμών και των προβλεπόμενων δαπανών. Πρέπει να κλείσει αυτό το χάσμα επίσης και σε σχέση με το πρόγραμμα COSME, το, οποίο περικόπηκε κατά 20%. Ε, με τις τωρινές προτάσεις το θα, πάμε, θα κατεβούμε στο μείον 10% αλλά δεν αρκεί αυτό. Προτείνω λοιπόν να γίνουν και άλλες κινήσεις για να μειωθεί και άλλο αυτό το χάσμα. Ως προς το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο οποίο δόθηκαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να έχουμε ένα σαφές κονδύλιο στον προϋπολογισμό, το το οποίο να πηγαίνει σε αυτό το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο ε, και για, την, ε, ε, για το Intelligent Energy Europe έχουμε την εμπειρία από το παρελθόν και τις εξοικονομήσεις που σημειώθηκαν και αφού ήταν μια ευνοϊκή εμπειρία νομίζω πρέπει να το διατηρήσουμε. Σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, ορισμένοι συνάδελφοι έχουν υποβάλει 7 συνολικά προτάσεις. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έχει στείλει την αξιολόγησή της για τις προτάσεις αυτές. Ε, αύριο υποτίθεται ότι θα έρθουν οι αξιολογήσεις αυτές. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρακτική να αναμένουμε την αξιολόγηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το λόγο αυτό δεν είμαι σε θέση τώρα να σας ε, πω κατά πόσο οι προτάσεις των συναδέλφων θα τύχουν της υποστήριξης ή της έγκρισης της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφος Ρουμπίκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Μπουτικόφερ. Είναι όντως δύσκολα τα προγράμματα αυτά να τα διαχειριστεί κανεί και αν δεν κανείς και το δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2007-2013 και το 2014 στο 20, το Συμβούλιο έχει μειώσει κατά 3,4% τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μέχρι το 2020 λοιπόν γίνονται πολύ μεγάλες περικοπές. Ε, βέβαια στα κράτη-μέλη δεν τη βλέπει κανείς αυτή την τάση και αναρωτιέμαι γιατί. Γι' αυτό νομίζω ότι το σχέδιο που έχουμε πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά, ας πούμε και την, τον εμπλουτισμό του ορίζοντα 2020, αν δούμε τι έχει προσθεθεί εκεί και τι πρέπει να καταβληθεί επιπλέον ε, ως δαπάνες, ε, δεν σημαίνει, ε, δεν αποτελεί ούτε δεν αποτελεί κατά ανάγκη αύξηση. Μιλούμε για τρία δις εκ των οποίων τα δύο επιστράφηκαν. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια θετική προσέγγιση. Υπάρχει και η πρωτοβουλία αυτή του front-loading. υπάρχει το Erasmus, κάποια μικρά ποσά έχουν προωθηθεί, έχουν αλλάξει η γραμμή, υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία έχει συμπληρωθεί για την, ε, για την διασύνδεση των ε, ενεργειών και με την ανάληψη ευθύνης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ταμείο Επενδύσεων. Εκεί μιλούμε για 10 δις επιπλέον και το, ένα, και το Ταμείο θα λάβει επιπλέον 1 δις. Ε, επίσης, τα δάνεια και εγγύσεις για τις μικρομεσαίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύ ισχυρό μοχλό πίεσης. Μιλούμε για 120 δις ευρώ. Με έναν πολλαπλασιαστή 1 έως 5 ή 1 έως 10. Μιλούμε δηλαδή για ένα εκατομμύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν για κάθε ε, νέο ε, εργαζόμενο να έχουμε μια εγγύηση 10.000 ευρώ, έτσι ώστε να υπάρξει μια κινητοποίηση σε ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα μπορούσαμε επίσης να εξεύρουμε και άλλους τρόπους, ας πούμε χρηματοδότηση εξαγωγών, ε, εγγυήσεις ε, αποδόσεων. Ε, θα μπορούσαμε όντως να βοηθήσουμε έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πολλές φορές δεν έχουν από μόνες τους το ίδιο κεφάλαιο. Πρέπει λοιπόν να το παρακολουθήσουμε στενά. Ξέρω βεβαίω ότι μπορώ να πιστεύω τον εισηγητή, θα το παρακολουθήσει στενά για να δούμε όντω ε, κατά πόσο είναι ή δεν είναι επαρκή τα συγκεκριμένα ποσά και νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε ένα συγκεκριμένο ε, θέμα ως κεντρικό άξονα έτσι ώστε να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τα λοιπά, ε, καλή επιτυχία στον ε, εισηγητή και καλή δύναμη στις διαπραγματεύσεις. Έλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορούμε να το συζητήσουμε στο και σύντομα το θέμα αυτό. Για την συζήτηση αυτή για τον, 2000, ε, για τον ορίζοντα 2020. να πω κάτι. Ε, για τα νούμερα. Η Κομισιόν έχει βάλει εδώ πέρα ένα αριθμό για τον ε, ορίζοντα 2020 ε, για ένα 20%. Είναι λάθος αυτό. Είναι μάλιστα κενό. Αν δούμε τους, τους, τους αριθμούς, το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και την Ευρατών έχουμε 59,2 δις. Αν δούμε τους αριθμούς του 2013, τότε βασιζόμαστε στις τιμές του 2011. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά βέβαια. Είμαστε στα 77,7 δις. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο λοιπόν συνδυάζει τα 77,78 δις και έχουμε και έναν ε, έναν προπολογισμό 70,2. Δηλαδή ε, μιλούμε για 10% περίπου, 9-10%. Ε, ναι, Δεν είναι απλά μαθηματικά αυτό, είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που μίλησε για το θέμα του front loading. Το 2014 θα είμαστε κάτω από, τους, ε, από τα όρια του 2013. Και αυτό δεν έχει, δεν έχει γίνει ποτέ από τότε που ξεκίνησαν τα προγράμματα έρευνα στην Ευρώπη. Και όλοι μιλούν κάθε φορά για καινοτομία, το οποίο το έχουμε συζητήσει και εμείς για την εκβιομηχάνηση, το ξαναείπαμε. Θα πρέπει λοιπόν τουλάχιστον να καταφέρουμε για τον ορίζοντα να μην βγει τελείως από την δυνατότητα ευελιξίας. Υπάρχουν κάποια κενά. Ε, τώρα δεν είναι στην ε, ευελιξία ο ορίζοντας, γι' αυτό χαίρομαι που ο εισηγητής ε, θέτει το θέμα αυτό του front-loading. Γιατί είμαστε και βεβαίως είναι τρέλα σε μια τέτοια κρίση να μειώσουμε τις επενδύσεις για την καινοτομία. Τα, τελευταία, τα επόμενα δύο χρόνια πρέπει να έχουμε επαρκή κονδύλια ακόμα και στο μειωμένο οικονομικό πλαίσιο που βρισκόμαστε, για να για να μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσει στην κοινοτομία, όχι να δημιουργήσουμε τώρα προβλήματα τα οποία θα φανούν σε 4-5 χρόνια. Πρέπει να δείξουμε και ένα μήνυμα και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και ένα προ τι προς τις ε, διεθνείς Επίσης, η επανεισρωή των κονδυλίων στον προπολογισμό. Έχουμε κάνει πολύ κουραστικέ διαπραγματεύσει προ αυτό και θα πρέπει να συμπληρωθεί οι, επιστροφέ στον προϋπολογισμό θα πρέπει να βγουν από τον ορίζοντα ακόμα και όταν πάρουμε πίσω τα χρήματα. Αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα που συζητείτε έχει οδηγηθεί τελικά σε, έχει μετατραπεί σε κοινό γράμμα. Σε κοινό γράμμα γιατί ούτως ή άλλως όλα τα χρήματα που επιστρέφουν επιστρέφουν στο γενικό προϋπολογισμό. Οπότε είναι καρικατούρα αυτό που έχουν, που έχουν προτείνει οι ηγέτες ε, κρατών και κυβερνήσεων. Στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να μπορούν ε, τα, ε, τα κονδύλια που δεν χρησιμοποιούνται να επιστρέφουν εκεί, εκεί από όπου δεν χρησιμοποιήθηκαν, όχι στο γενικό προϋπολογισμό. Γιατί μέχρι τώρα πηγαίνουν όλα στο γενικό προπολογισμό. Η ρητορική λοιπόν ε, δεν κατοπτρίζει αυτό που γίνεται τελικά στις διαπραγματεύσεις. Παρόλα... Ωραία. Ο λόγος τώρα στον εισηγητή για να απαντήσει, παρακαλώ. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Ρούμπικ και τον κύριο Έλερ. Τον ε, προπολογισμό που έχει δεχτεί το Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε να τον αποτρέψουμε, να... ακόμα και αν μας πονάει, αν μας ενοχλεί. Δεν έχουμε επαρκή κονδύλια. Απλώς προσπαθούμε να κάνουμε τα πικρά γλυκά. Έτσι πρέπει να το πω. Αν συγκρίνουμε τα νούμερα, ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7, 2013, 10 δις, ορίζοντας 2020-2014, 8,8. Ακόμα κι αν κάνουμε με το front loading, αν βάλουμε 200 εκατομμύρια παραπάνω, πάλι δεν λύνεται το πρόβλημά μας. Ακόμα και αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα, όλα τα περιθώρια που έχουμε, δηλαδή περίπου 400 εκατομμύρια και ακόμα και χρησιμοποιήσουμε όλο το περιθώριο από την ευελιξία, πάλι 400 ε, εκατομμύρια είναι, πάλι δεν καταλήγουμε στο status quo. Και το αν θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα περιθώρια βέβαια είναι άλλο θέμα. Οπότε συμφωνώ με αυτό που λένε οι συνάδελφοι. Το ερώτημα απλώς είναι αν αυτή η Επιτροπή, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, μπορεί να βρει κάποια μέσα, όχι μόνο για να παραπονεθεί, αλλά για να μπορέσει να ε, προειδεάσει ή να επηρεάσει λίγο τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Βεβαίως θα δεχτώ, δέχομαι όλα όσα είπατε και θα τα έχω υπόψη μου. Ωραία, ευχαριστώ. Να υπενθυμίσω σε όλους τους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την κατάσταση των τροπολογιών είναι 3η 20 Αυγούστου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα... Την γνωμοδότηση του κυρίου Οντή ε, για το σημείο 19 θα μεταφέρουμε τη συζήτηση ε, για το απόγευμα ε, μετά από την παρέμβαση των Υπουργών. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χίμπνερ, το σημείο 17 εννοούσε η Πρόεδρος και να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ντί για την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προς το παρόν δεν υπάρχει έγγραφο. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για μια γνωμοδότηση την οποία θα κάνουμε για την τεχνολογική και βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Πρόκειται για κάτι λίγο πιο ιδιαίτερης φύσεως, ε, μία έκθεση ε, της Υποεπιτροπής Άμυνας και ζητά τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την οποία αποφάσισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. να συγκαλέσει το Δεκέμβριο για το θέμα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Πρόκειται για ένα πιο ιδιαίτερο ζήτημα. Δεν είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας την οποία υποβάλλουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αποτελέσει κίνητρο για νομοθετικές προτάσεις. Είναι μια έκθεση ε, την οποία υποβάλλουμε προκειμένου να δούμε λίγο ε, εάν οι ιδέες των Ευρωβουλευτών ενδιαφέρουν τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για την άμυνα των χωρών τους. Το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ περιορισμένο, διότι μετά από αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα μιλήσουμε με τους ε, εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες και θα υποβάλω ένα σχέδιο γνωμοδότησης ε, προς μετάφραση, το οποίο θα συζητήσουμε το Σεπτέμβριο με ψηφοφορία ε, στην Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Νοέμβριο. Υπάρχει μια μελέτη την οποία σας προτείνω να διαβάσετε της ε, ε, νομικής ομάδας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Άμυνας και από τα στοιχεία που μου έχουν δοθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία σίγουρα θα δεχτεί να μας πει δύο λόγια, θα πρέπει να κάνει μια ανακοίνωση στα μέσα Ιουλίου για τον τομέα οι ευρωπαϊκές αγορές ε, της ε, ε, βιομηχανίας άμυνας εκπροσωπούν 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι αμερικανικές βιομηχανίες έχουν ένα τμήμα της αγοράς περίπου το 50% και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε περίπου το 20%. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι κατά πόσον η ευρωπαϊκή ζήτηση είναι επαρκής ώστε να μπορέσει να τροφοδοτήσει μια βασική ε, ευρωπαϊκή άμονα, αν ε, είναι προσαρμοσμένες οι ανάγκες μας ε, στα αιτήματα της αγοράς και αν καλύπτει η προσφορά τη ζήτηση και αν και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας αυτής της αγοράς. Θα πρέπει επίσης να δούμε ποιοι είναι οι παράγοντες της αγοράς, οι διεθνείς παράγοντες και να δούμε επίσης και αν όπως κάνουμε τώρα, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε ακόμα περισσότερο, να αναπτύξουμε κατάλληλα συστήματα άμυνας, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι προσβάσιμα μόνο από συγκεκριμένε βιομηχανικές ομάδες που μπορούν να αναλάβουν κινδύνους και να εξετάσουν το πόσο ευαίσθητη είναι αυτή η τομή. Υπάρχει και ανάγκη για συγκεκριμένε τεχνολογικές δεξιότητες, ε, επίσης ε, κατάλληλες ε, οικονομικές γνώσεις και φυσικά η κατάλληλη πρακτική στις διεθνείς αγορές. Αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ADS, οι Ταλής, οι Φινμεκάνικα ε, έχουν κατάλληλα συστήματα και έχουν και δίκτυα υπεργολάβων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε θέματα αεροπλάνων, ε, ε, σκαφών, παραδοσιακής άμυνας, πυράβλων και το καθεξής. Και σήμερα διαπιστώνουμε, και με αυτό θα ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε για την πρώτη εισαγωγή μου εδώ, με τη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει μία στρατιωτική αλληλεγγύη από πλευράς όλων των κρατών για την προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών. Πρόκειται για μία δυνατότητα στρατιωτικής αλληλεγγύης βάση του σχετικού άρθρου της συνθήκης ε, ε, αντίστοιχη με ε, το άρθρο που υπάρχει στην Συμφωνία του ΝΑΤΟ και μέχρι τώρα αυτό που βλέπαμε ότι όποτε υπήρχε κατοχή εδαφών, ε, η συνεισφορά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας ήταν πολύ σημαντική. Αρχίσαμε λοιπόν να αναρωτιόμαστε στον περίπλοκο κόσμο του σήμερα πώς μπορούμε να οργανωθούμε από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα οργανώσουμε τη βιομηχανική βάση άμυνας ώστε να υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση, ώστε να γίνουμε και οι καλύτεροι σε θέματα ε, τεχνολογίας και επιστήμης, τα οποία θα συνεισφέρουν μεν, ε, αλλά ταυτόχρονα θα, πώς θα έχουμε και τα κατάλληλα υλικά για να έχουμε μια κατάλληλη ε, βιομηχανική βάση άμυνας. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική βοήθεια, γνωρίζουμε ότι στις δύσκολες πολιτικές συμφωνίες τις οποίες καταλήξαμε για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν μπορούμε να διαθέσουμε κανένα κονδύλιο προς το παρόν. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα της ρήτρα αναθεώρησης του 2016 η οποία πιστεύω, εάν βρούμε φυσικά και την κατάλληλη πλειοψηφία για το θέμα αυτό, ε, θα μας επιτρέψει να θέσουμε το θέμα αυτό προς συζήτηση για τις ευρωεκλογέ του 2014. Θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορεί να φύγει και το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα βρεθούμε ενώπιον μιας νέας πραγματικότητας και θα πρέπει να εξετάσουμε τι θα γίνει επί τη βάση των εγγράφων τα οποία ε, ξεκινούμε σιγά σιγά σποραδικά να ετοιμάζουμε για να δούμε αν η ιδέα της ύπαρξης μιας ε, βιομηχανικής βάσης άμυνας ε, βρίσκει σύμφωνος και τους πολιτικούς ηθήνοντες και αν θα μπορούμε να έχουμε και την κατάλληλη πλειοψηφία ε, διότι η Ευρωπαϊκή Άμεση να πρέπει να διαδραματίσει ένα επιπλέον ρόλο. Βέβαια είναι περιορισμένοι οι προπολογισμοί των κρατών μελών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν μπορούμε να έχουμε αμοιβαία συνεργασία ώστε να μπορέσουμε εμεί ω Ευρωπαίοι να είμαστε οι καλύτεροι σε επιστημονικό, τεχνικό επίπεδο και για να υποστηρίξουμε και τη βιομηχανική μα βάση. Αυτά λοιπόν, δύο λόγια, προσκέψη και συζήτηση κυρία Πρόεδρε. Αδειμονώ να μάθω και τις απόψεις ε, των υπολείπων για τα θέματα αυτά τα στρατιωτικά θέματα, τα θέματα άμυνας και ασφαλείας ε, θα τα καλύψει η Επιτροπή Άμυνας και εμείς από πλευράς Επιτροπής μας θα ασχοληθούμε ε, με τα θέματα της επιστημονικής έρευνας, τα τεχνολογικά και όλα τα βιομηχανικά στοιχεία και σε αυτό θα πρέπει να ε, επικεντρωθούμε και φυσικά και στην ενέργεια. Ο κύριος Γκέρεκ παρακαλώ. Γκέρεκ, πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ το εξής. Πρέπει να καθορίσουμε με μεγάλη σαφήνεια ποιος είναι ο στόχος μας. Ίσως να είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα κοινό σύστημα άμυνας, αμυντικής βιομηχανίας, αλλά πολύ απέχουμε ακόμη από αυτό. Τα εθνικά συστήματα ε, είναι προστατευμένα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους και είναι πολύ ερμητικά υπό μία έννοια. Κάθε χώρα έχει το δικό της αδιαπέρατο, αδιαπέραστο σύστημα, ε, στεγανό σύστημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ε, η κληρονομιά της ε, αμυντικής βιομηχανίας από τα δύο μεγάλα αντίπαλα στρατόπεδα ε, είχαμε το σύμφωνο της Βαρσοβίας από τη μία πλευρά και ένα εντελώς, μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από την άλλη πλευρά και αυτά τα δύο πρέπει κάπως να ενοποιηθούν, να ομογενοποιηθούν γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές όσο αφορά την τεχνολογία και τις προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό Ιδίω όσο αφορά τα, τις προδιαγραφές, τα πρότυπα, χρειαζόμαστε συνεργασία. Ας πάρουμε τα πυρομαχικά. Τους, ε, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις νομοθεσίες μας να συγκλίνουν κατά κάποιο τρόπο. Ε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την προμήθεια των πυρομαχικών. Ε, χρειάζεται ομογενοποίηση των προτύπων. Ένα, άλλο θέμα τώρα πάνω στο οποίο εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές. Πολύ χρήσιμο νομίζω θα ήταν να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες συνέργειες ή να τις δημιουργήσουμε, να, βρούμε, να αναζητήσουμε το κοινό έδαφος. Και ακόμα και αυτό το 20% αυτών των 350 δισεκατομμυρίων αποτελούν μια πολύ καλή αφετηρία. Ας το κάνουμε αυτό στην ε, ε, αεροπορία, στην αμυντική αεροπορία, αλλά και στα τεθωρακισμένα ε, οχήματα και σε άλλα οχήματα, γιατί όχι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε αυτό πιο εκτεταμένα. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια συνάντηση. Ε, ο κύριος Οντί θα οργανώσει μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Πουτικόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας που γράφει ο κύριος Γκάλερ για την ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ. Αλλά εγώ μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει τίποτα από τον ίδιο. Τι ακριβώς δηλαδή θέλει να κάνει με αυτή την έκθεση. Οπότε ε, απλώς να υποθέτω μπορώ. Και άκουσα ότι αύριο θα γίνει η συνάντηση των σκιωδών. Ε, τη βάση τι θα γίνει αυτό. Ε, Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί τα προβλήματα που αναφέρονται είναι παμπάλαια. Οι ελλείψεις ε, σε επίπεδο ικανοτήτων και σε ό,τι αφορά την ΚΕΠΑ και σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Ε, εδώ και 14 χρόνια τα ξέρουμε από τον πόλεμο στο Κόσοβο. Ε, μετά το έδειξαν και οι διάφορες δραστηριοποιήσεις στην ε, Λιβύη. Η δυσκολία νομίζω βρίσκεται κυρίως στο ότι τα κράτη-μέλη κρατιούνται σε μια αναχρονιστική αμυντική βιομηχανία. Μιλούμε για διεφθαρμένες ηγεσίε, μιλάμε και για έναν εθνικιστικά περιορισμένο ορίζοντα δυνατοτήτων. Ε, με τα χρήματα που, μπορούσε, που δίνονται σε αυτόν τον, τον κλάδο της άμυνας θα μπορούσε κανείς να έχει κάνει θαύματα εάν ήταν διαφορετικές προοπτικές και αν ήταν και διαφορετική η διαχείρισή τους. Δεν βλέπω λοιπόν πώς αυτό θα αλλάξει άμεσα αν δείτε τι γίνεται και στο pooling and sharing ας πούμε. Μιλούμε για 300 προτάσεις που έχει κάνει ο ίδιος ο στρατιωτικός κλάδος. 11 έχουμε συμπεριλάβει. Ε, καταλαβαίνετε, λείπει η βούληση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, θα πρέπει να, πάμε, να είμαστε τόσο ακραίοι, να πάμε τόσο μακριά και να πούμε το άρθρο 346, μήπως πρέπει να το διαγράψουμε, το οποίο είναι αυτό που εγγυάται στα κράτη-μέλη ότι λόγω εθνικής ασφάλειας ή τέλος πάντων κάτω από αυτό το μανδύα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με την αντιμετική τους βιομηχανία. Αν παραμείνουμε σε αυτό το, άρθρο, καμιά ε, Ευρώπη δεν θα μπορέσει να φτάσει σε αποτελεσματική χρήση των πόρων και σε μια σωστή αμυντική βιομηχανία και βεβαίως έτσι δεν θα κλείσουν και τα κενά που υπάρχουν στην βιομηχανία. Γι' αυτό νομίζω ότι Καλό είναι που, έχουμε, που κάνει ο κύριος Γκάλερ αυτή την ε, έκθεση, γιατί ξέρω ότι είναι καυτό το θέμα, αλλά αν έχει νόημα να κάνει κανείς μια τέτοια έκθεση, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος, να μην αμβλύνει απλώς κάποιες γωνίες ή να λέει έτσι περί διαγραμμάτων τι πρόκειται να κάνει. Θέλουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο που θα ανοίγει ένα νέο ορίζοντα, γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα παραμείνουμε πίσω από αυτά που ήδη έχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ταζενόσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κύριος Σοντέ. Ε, πριν από δύο χρόνια ήμουν εισηγητής ε, για την βιομηχανία της άμυνας και τότε, πριν από δύο χρόνια, αντιλήφθηκα πόσο περίπλοκο είναι αυτό το σύστημα της βιομηχανίας άμυνας. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για ανοιχτή αγορά, όπως είπαν οι συναδελφοί. Πρόκειται για μια πολύ εξειδικευμένη αγορά, ιδίως ε, σε θέματα εθνικών διαδικασιών και ταυτόχρονα είναι και μια τεράστια βιομηχανία. που φυσικά έχει και αντίστοιχο οικονομικό αντίκτυπο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δούμε πώς θα πρέπει να ασχοληθούμε με την βιομηχανία της άμυνας, ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με πολύ περίπλοκα πράγματα, διότι κάθε κράτος μέλος εγκρίνει διαφορετικά πράγματα και υπάρχουν και αποκλίνουσες θέσεις. Συμφωνώ απολύτως ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Προφανώς και θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα πρέπει να δράσουμε στον τομέα αυτό. η επιστήμη και η έρευνα έχουν πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν στον τομέα, διότι η τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας είναι ε, πάρα πολύ μεγάλη και η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να αποτελέσουν σύνδεσμο για αυτήν την τόσο κατακαιρματισμένη αγορά της ε, βιομηχανίας της άμυνας. Με τα χαράς ε, να συνεργαστώ με τον κύριο Ντί. Εδώ και δύο χρόνια ε, είχαμε συζητήσει για το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, αλλά είμαι διατεθειμένος να συνεισφέρω όσο περισσότερο μπορώ με τις ιδέες μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριο Σέλλερ. Τέθηκε το ερώτημα για το πώς διαχειρίζεται κανείς το θέμα αυτό, ε, τι μπορούσε να κάνει ο κύριος Γκάλερ. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το δούμε στα πλαίσια και των όσων έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Έχουμε πολλές ε, εκθέσεις για τις ε, δυνατότητες των στρατιωτικών δυνάμεων της ε, Ένωσης και σε ό,τι αφορά την αμυντική πολιτική. Πάντα υπάρχει ένα κεφάλαιο για την βιομηχανική πολιτική. Είναι σημαντικό το ότι το θέμα αυτό είναι κοινό για όλους, ακριβώς λόγω της ευρωπαϊκής του διάστασης. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία θα βασίζεται σε ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι ώστε να λύσει τα διάφορα διλήμματα που υπάρχουν η αρμοδιότητα είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης είναι και επιθυμητό να γίνει κάτι τέτοιο. Οπότε το ερώτημα θα πρέπει να είναι, θα συμφωνήσουμε να προχωρήσουμε από κοινού ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ως προς τον κλάδο αυτό, ως προς τον τομέα αυτό. Και θα πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για τις ευρωπαϊκές δυνατότητες, όχι για τις, ευρωπα... για τις εθνικές δυνατότητες. Γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια βάση συζήτησης. Έχουμε την κοινή πολιτική άμυνας. Ε, λαμβάνονται αποφάσεις, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε δυνατότητες. Ας πούμε, ε, ολοκλήρωση, επικοινωνία, αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε και σε ό,τι αφορά την επιχειρησιακή του πτυχή, αλλά και την πολιτική του πτυχή. Καθώς επίσης και λόγω της αναγκαιότητας που υπάρχει να υπάρξει σε αυτό τον τομέα μια ιστορική αγορά. Νομίζω λοιπόν ότι από την πλευρά της δομής θα πρέπει να είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, πώς θα δραστηριοποιηθούμε και στα πλαίσια των ε, αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί. Το θέμα δεν είναι απλώς να κοιτάμε από την, ε, ε, τα κράτη-μέλη να κοιτούν ε, την Ευρώπη για να τους λύσει το πρόβλημα, τώρα που βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης, αλλά πρέπει το Κοινοβούλιο και γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε μια εθνική προσέγγιση. Ευχαριστώ, συνάδελφο Σοντή. Έχετε το λόγο. Κύριο Σοντή. Ε, ε, σχόλιο εκτός μικροφώνου. Α, ναι, ναι, είναι η σειρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθήσαμε να την παρακάμψουμε. Θέλετε να πείτε κάτι εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Okay, Εντάξει, τάχιστα παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα απλά να επιβεβαιώσω αυτό που υπόθηκε για την επερχόμενη ανακοίνωση που προετοιμάζει η Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Αληθεύει. Η ανακοίνωση αυτή θα εγκριθεί είτε στις 24 είτε στις 25 Ιουλίου. Το έγγραφο αυτό θα συζητηθεί σε μια άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου στη διάρκεια της Προεδρίας της Λιθουανίας Υπάρχει και η δεύτερη έκθεση που προετοιμάζεται από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή στο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και θα ασχολείται με το θέμα της ικανότητας ε, και θα συμπληρώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Οντί, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων ακριβώς αναδεικνύει ε, το περίπλοκο του θέματος. Νομίζω ότι η πολιτική ανάγνωση του 21ου αιώνα ε, δεν μπορεί να είναι ίδια με την ανάγνωση του 20ου αιώνα. Όλος, ο καθένας το καταλαβαίνει αυτό. Σημερίζομαι τις ανησυχίες των βουλευτών ε, για τις εθνικές νομοθεσίες. Ε, τα στρατιωτικά θέματα έχουν μια έντονη εθνική συνιστόσα. Ε, υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αρχηγών κρατών πάνω σε αυτό. Η πρόταση που σας κάνω εγώ είναι να έχουμε ένα έγγραφο προβληματισμού για να δούμε τι πολιτικές πλειοψηφίες μπορούμε να συγκεντρώσουμε, ποια θα είναι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, η οποία θα παραδοθεί στους αρχηγούς κρατών σε συνδυασμό φυσικά και σε διαβούλευση με την Επιτροπή Άμυνας. Ε, και βέβαια θα αποφανθούν και οι πολίτες ε, ε, θα δώσουν την ετοιμιγορία τους ε, έχοντας γνώση τη γνωμοδότηση αυτή. Ε, έχουμε την ευρωπαϊκή γεωγραφία του 21ου αιώνα η οποία δεν μπορεί να είναι ίδια με αυτό που συνέβη στο παρελθόν ούτε καν στη διάρκεια της μεταβατικής κατάστασης που περνάμε τώρα. Ε, βέβαια δεν πρόκειται ούτε του 2013 ούτε του 2014 να το ρυθμίσουμε το θέμα. Είναι πιο μακρόπνο, πιο μακροπρόθεσμο. Εάν αποφασίσουν από κοινού οι αρχηγοί κρατών να κάνουν κάτι ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους μεγαλύτερους στρατούς της Ευρώπης, ο τελευταίος στρατός της Ευρώπης αν θέλετε. Αν όμως ε, αφήσουν ε, τους υπόλοιπους στο στρατιωτικό πεδίο θα δούμε τι θα γίνει. ως για το άρθρο 346. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το αλλάξουμε. Δεν είμαστε ομοσπονδία. Είμαστε ένα συνασπισμός κρατών. Τα κράτη είναι Εθνικός κυρίαρχα. Ε, θα κάνουν αυτό που θέλουν. Θα μείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα φύγουν, θα εθνικοποιήσουν ε, κάποιες επιχειρήσεις. Δεν θα τις ε, εθνικοποιήσουν. Έχουν τις δικές τους ανησυχίες του εθνικού συμφέροντος. Είναι γενικότερο το θέμα. Το θέμα είναι εάν στον τομέα ενδεχομένως της άμυνας. Ε, ε, αν μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση, αν υπάρχει κάποιος ευρωπαϊκός δρόμος. Αυτό είναι το θέμα πάνω στο οποίο εργαζόμαστε αύριο, στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών που σας προτείνω. Δεν θα υπάρξει έγγραφο, δεν θα υπάρξει κείμενο. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε βαθύτερα σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων εγώ θα ετοιμάσω κάτι, θα το υποβάλω για μετάφραση και θα δω με τους φίλους μας, ε, με τον φίλο και βουλευτή Γκαλέγα, ε, θα δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς για να δώσουμε και ένα μήνυμα στους αρχηγούς των κρατών.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 θέλουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, οπότε την έκθεση για τον, 2000, ε, για τον 2020 ίσως να πρέπει να τη δούμε το Σεπτέμβρη. Δεν, λέω, δεν το λέω γιατί δεν υπάρχει θέληση από τους ε, συναδέλφους να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους, αλλά θα είναι πραγματικά ε, σε πέντε λεπτά, θα είναι αστείο σε πέντε λεπτά να προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε για ένα κείμενο που τρέχει εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο. Ίσως λοιπόν θα μπορούσατε να ενημερώσετε και τους άλλους συναδέλφους, γιατί ε, τώρα και χωρίς ε, διερμηνία και έχουμε και τρία λεπτά στη διάθεσή μας, δεν γίνεται να ενημερωθούμε εντελεχώς. Δεν λέω γιατί δεν θέλετε να το πράξετε, λέω γιατί δεν γίνεται για ένα τέτοιο θέμα πέντε λεπτά να αφιερώσουμε μόνο για να το δούμε. Ε, Πρώτον λοιπόν, η πρόταση του κυρίου Έλερ και της κυρίας Μαντουρέλ μου φαίνεται λογική να τα συζητήσουμε στο, το Σεπτέμβριο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τερέζα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, εγώ δεν έχω καμία ένσταση. Συμφωνώ με αυτό που προτείνει ο συνάδελφος Έλερ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε σήμερα μια σύντομη ενημέρωση διότι θα υπάρξει συζήτηση στην Επιτροπή και ψηφοφορία το Σεπτέμβριο. Πρέπει να ψηφίσουμε λοιπόν. Υπάρχουν δύο λύσεις, οποιαδήποτε και αν επιλέξετε καλή είναι. Ναι, σίγουρα όχι τώρα. Θα το δούμε με τη γραμματεία και θα προσπαθήσουμε να βρούμε λίγο χρόνο ώστε να γίνει μια ενημέρωση. Όχι αυτή τη στιγμή διότι δεν είναι δυνατόν. Τώρα θα ήθελα να διορθώσω ένα λάθος που έκανα εγώ διότι δεν είναι 2 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα γίνει η συζήτηση για την γνωμοδότηση του κυρίου Οντή και η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών δεν έχει ακόμα καθοριστεί. Θα ήθελα επίσης ε, να σας ενημερώσω ε, για την συνεδρίαση των συντονιστών εχθές. Καταλήξαμε σε συμφωνία μεταξύ των συντονιστών για τη διαδικασία της Επιτροπής Ήτρε για τις κατεξουσιοδότησης πράξης και αποφασίστηκε ότι όταν 7 τακτικά μέλη που προέρχονται από διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν ένσταση, θα επιτρέπεται να εγγραφεί το σημείο στην ημερήσια διάταξη ή όταν ε, οι συντονιστές ξεκινούν τη διαδικασία θα μας επιτρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία για συζήτηση μιας κατεξουσιοδότησης συμπράξης και στη συνέχεια ψηφοφορία. Αυτά έχουν διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους και επίσης ε, καθορίστηκε να αναλάβουν οι σοσιαλιστές το πρόγραμμα έρνικος και ε, δόθηκαν και τέσσερα εκθέσεις και ένα προφορικό ερώτημα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στους ε, συντονιστές. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε θα ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση εδώ και θα συνεχίσουμε στις 3. Έχουμε τους ε, δύο υπουργούς και κατόπιν την Επίτροπο μετά από κάποια θέματα άλλα. Ευχαριστώ. Τα λέμε στη συνέχεια.